Chers collègues, euh, bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας προτείνω να ξεκινήσουμε. Ελπίζω ο κύριος Όρη να γυρίσει να με κοιτάξει. Να μου έχει την πλάτη γυρισμένη. Ε, c'est notre première réunion de euh, l'année 2011, donc... Είναι η πρώτη συνεδρίαση του 2011 και θα ήθελα επί της να σας ευχηθώ κάθε ευτυχία και προσωπική ευτυχία και επαγγελματικές επιτυχίες και θα μπορέσουμε να το πούμε αύριο περισσότερο ανεπίσημα. Για την μείσια διάταξη έχουμε δύο μικρές τροποποιήσεις για το θέμα της στρατηγικής και της ενσωμάτωσης των Ρωμά στο σημείο 11 θα συζητηθεί μετά το σημείο 12. Και το σημείο 13, η έκθεση Κοφεράτη για τη σημερινή κατάσταση και τις μελλοντικέ συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαφορετικών ταμείων θα ε, πάει στη θέση του σημείου 26 και το σημείο 26 το σημείο του 13. Το σημείο 11 λοιπόν θα γίνει σημείο 13 και το σημείο το τωρινό 13 θα αντικατασταθεί με το σημείο 26 και αντιστρόφως. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Και έχουμε διάφορες εκθέσεις ε, για τις συναντήσεις ε, στη Θεσσαλονίκη και για επισκέψεις σε διαφόρους οργανισμούς. Έχετε λάβει και τα πρακτικά της συνεδρίασης στο Τωρίνο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό κατάρτισης. Έχετε λάβει και τα πρακτικά της ε, αντιπροσωπείας στην αποστολή της στην Ουγγαρία. Επίσης θα βρείτε το σημείο που μας έχει προετοιμάσει η Γραμματεία και ευχαριστούμε πολύ τη Γραμματεία για αυτό το σύντομο σημείωμα. Σχετικά με την ακρόαση της Επιτροπής για ένα κατάλληλο και βιώσιμο σύστημα συνταξιοδότησης στην Ευρώπη. Όλα αυτά σε σχέση με την έκθεση Όιμεν ΡΟΙΤΑΝ. Επίσης έχετε πρακτικά από μία ακρόαση για το μέσο μικροχρηματοδότησης. Επίσης αύριο θα λάβετε ένα σημείωμα για την αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης ε, η οποία υπόκειται σε μια σοβαρή αναδιάρθρωση και φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται όλοι οι συνάδελφοι. Θέλουμε να ξέρουμε πού βρίσκονται οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή και αυτοί με τους οποίους θα ερχόμαστε σε επαφή στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Έχετε τα πρακτικά της 22 Νοεμβρίου και της 1ης και 2 Δεκεμβρίου. Και αν έχετε παρατηρήσεις, παρακαλώ μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να μας τα υποβάλλετε. Διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνουν τα πρακτικά όσα έχουν. Περνάμε στο πρόγραμμα εργασιών των οργανισμών. Είναι σημαντική αυτή η παρουσίαση και για τους οργανισμούς αλλά και για μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο τη δουλειά ενός χρόνου να την παρουσιάσετε μέσα σε πέντε λεπτά, αλλά γνωρίζετε τις δυσκολίες ε, που υπάρχουν και γι' αυτό ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα δώσω το λόγο σε κάθε οργανισμό και στη συνέχεια θα αρχίσει η συζήτηση για όλους τους οργανισμούς από κοινού. Με βάση τη ημερήσια διάταξη, δίνουμε καταρχήν το λόγο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και καλή χρονιά σε όλους. Από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ένα από τα βασικά μας έργα για την περσινή χρονιά ήταν να συντονίζουμε όλους τους οργανισμούς στο ευρωπαϊκό σύστημα, 28 οργανισμούς δηλαδή συνολικά. Φαντάζομαι ότι θα έχετε τα έγγραφα σε διάφορες γλώσσες. Εδώ έχουμε μόνο τα βασικά σημεία που θα αναφέρω εγώ στην παρουσίασή μου. Τα βασικά σημεία καλύπτουν αυτό το οποίο έχουμε ως αποτέλεσμα από την προηγούμενη εκστρατεία μας για την αξιολόγηση κινδύνων. Ξεκινήσαμε πέρυσι μια δραστηριότητα για, την, για το εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου διαδραστικά, το ΟΙΡΑ. και ελπίζουμε ότι όχι μόνο για το 2011 αλλά για τα επόμενα 4-5 χρόνια θα έχουμε συνεχώς βελτιώσεις για το εργαλείο αυτό. Είναι εργαλεία που δίνουν στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα ε, να κάνουν την αξιολόγηση κινδύνου ε, στη γλώσσα τους και προσαρμοσμένο στι πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητε. Επίσης, δεύτερον, έχουμε την εκστρατεία για την υγεία στο χώρο εργασία ε, με βάση την ασφαλή συντήρηση και ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα. Τρίτη μελέτη είναι η Ευρωπαϊκή Έρευνα Επιχειρήσεων για νέους και αναδυόμενους κινδύνους. Επόμενο πρόγραμμά μας είναι τα, οι καλές πρακτικές και οι επιπτώσεις της ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στο Μπιλμπάου συνεχίζουμε με τα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά τη Συμφωνία για την Έδρα. Έχουμε κάνει πολλές ε, προσπάθειες και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε ε, τις προσπάθειες ε, ώστε να μην είμαστε σε αυτό το κτίριο για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη γιατί μπορεί να είναι ωραίο κτίριο αλλά είναι πανάκριβο. Πληρώνουμε ένα εκατομμύριο ενώ άλλοι οργανισμοί πληρώνουν ένα συμβολικό ποσό του ενός ευρώ το χρόνο συνδυάζουμε τις ε, διάφορες μονάδες για την αξιολόγηση κινδύνου και για το παρατηρητήριο, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την κατάσταση, αν και δεν έχουν αλλάξει πολλά επί της ουσίας. Αν δείτε τα όσα έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια, θα δείτε ότι πολλές χώρες έχουν προοδεύσει κατά πολύ στην ασφάλεια και υγεία, ενώ σε άλλες χώρες δεν είχαμε μεγάλη πρόοδο, είχαμε πολύ μικρή πρόοδο αυτή την διαφάνεια βλέπετε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που δείχνει ότι τα κράτη-μέλη που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχουν υποφελήθει περισσότερο και έχουν βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας περισσότερο σύμφωνα με την άποψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ήταν μια δημοσκόπηση. Το εργαλείο OIRA, το επιγραμμικό διαδραστικό εργαλείο ανάλυσης κινδύνου που σας ανέφερα, είναι κάτι που ξεκίνησε αρχικά στις κάτω χώρες και προσπαθούμε να το κάνουμε ένα γενικευμένο εργαλείο που θα χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε χώρα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις που δεν ξέρουν πώς να κάνουν αξιολόγηση κινδύνου. Αν δεν κάνει κανείς αξιολόγηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης, ε, ξεφεύγουν πολλά προβλήματα που έχουν σχέση με κινδύνους. Αυτό το εργαλείο βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορεί να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί και σε συσκευή PDA. Μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητε που είχαμε είναι η έρευνα επιχειρήσεων για νέους και αναδιόμενους κινδύνους. Συνεχίζεται η εργασία επί της λεπτομερούς αναλύσεως. Το χωρίσαμε σε περίοδους 2 ή 3 ετών και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά τη γνώμη των επιχειρήσεων. Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα είναι καταρχήν τα ατυχήματα, μυοσκελετικές διαταραχές και το στρες που οφείλεται στην εργασία. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου και τις επικίνδυνες ουσίες αλλά τα τρία πρώτα που σας ανέφερα είναι αυτά τα οποία αποτελούν την πηγή των περισσότερων απουσιών από την εργασία. Αν δούμε τις επιδόσεις των διαφόρων χωρών σε επίπεδο επιχείρησης, θέσαμε το ερώτημα αν υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη πολιτική, ένα σύστημα διαχείρισης ή πρόγραμμα δράσης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια μέσα στην επιχείρηση. Έχουμε πολλές θετικές απαντήσεις. Ε, τα καλύτερα στοιχεία τα παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχουν και χώρες που είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα για να δούμε τι γίνεται σε πρακτικό επίπεδο στις επιχειρήσεις. Σχετικά με τα νέα προβλήματα και το ρόλο του άγχους, του στρες που έχει σχέση με την εργασία, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, χώρες στις οποίες υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το άγχος και προσπαθούν να αναλάβουν δράση για να το αντιμετωπίσουν. Δεξιά βλέπετε ε, στο, στην εικόνα, στο δεξί σημείο βλέπετε τις χώρες που ανησυχούν και που λαμβάνουν μέτρα και τις χώρες που μπορεί να έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν έχουν αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσουν το στρες στο χώρο εργασίας. Μεγάλη σημαντική δραστηριότητα από το περσινό έτος ε, είναι η εκστρατεία για την ασφαλή συντήρηση. Η συντήρηση είναι μια δραστηριότητα που δεν είναι εύκολο να προγραμματιστεί γιατί πολλές φορές δεν είναι σταθερές οι συνθήκες και πολύ συχνά πρέπει να γίνεται η συντήρηση σε ε, απροσδόκητες συνθήκες και υπάρχουν ε, προβλήματα που σχετίζονται με τα ατυχήματα και με μειοσκελετικές διαταραχές που έχουν σχέση με τη συντήρηση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία που οργανώσαμε μέχρι τώρα, όχι διότι ήταν πολύ δαπανηρή, αλλά διότι κατορθώσαμε να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη καθώς και τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες ΕΖΕΣ να διοργανώσουν αυτή την εκστρατεία στη γλώσσα της η κάθε χώρα. Είχαμε μεγάλη παραγωγή στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, πάνω από 2 εκατομμύρια ε, είναι ο αριθμός των προϊόντων που θέσαμε σε κυκλοφορία. Συμπεριλαμβάνονται φυλάδια, ενημερωτικά δελτία, γελιογραφίες κλπ. Κάποια στοιχεία τώρα για το που βρισκόμαστε σήμερα και τι θα γίνει στο μέλλον. Πρόσφατα οργανώσαμε μια σχετικά μεγάλη μελέτη για το κόστος των οδηγιών για την ασφάλεια και την υγεία. Παρουσιάστηκε πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η μελέτη. Είναι μια μελέτη που έγινε σχετικά γρήγορα, αλλά είναι μια μελέτη που αντικατοπτρίζει αρκετά καλά τις απόψεις των διαφόρων φορέων και των ενδιαφερομένων στον χώρο εργασίας. αντί να μειώσουμε τα στοιχεία της αξιολόγησης κινδύνου, όπως είχε προταθεί από την έκθεση Στόιμπερ στο παρελθόν, η αντίδραση ήταν ότι δεν έπρεπε να μειωθεί αυτή η απέτηση. Καταρχήν διότι δεν θα εξοικονομούσαμε πολλά χρήματα και δεύτερον διότι θα επιδεινώνονταν οι συνθήκες στο χώρο εργασίας αν γινόταν κάτι τέτοιο. Αν δείτε τι έγινε στα πλαίσια της κρίσης, βλέπουμε ότι μειώθηκαν τα ατυχήματα γιατί είχαμε ε, μικρότερο ποσοστό κατασκευών, λιγότερες δραστηριότητες. Επομένως, τα ατυχήματα μειώθηκαν γιατί περιορίστηκαν οι δραστηριότητες που δημιουργούσαν τα περισσότερα ατυχήματα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ε, επιπτώσεις ε, στην επιδείνωση των συνθήκων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη διάσκεψη κορυφής είχαμε υπουργούς από την ε, Σουηδία και από την Ισπανία και ο Σουηδός υπουργός είπε ότι ένας στους τρεις εργαζομένους είναι εκτός εργασίας, όχι λόγω ανεργίας, αλλά λόγω μόνιμης αναπηρίας ή ασθένειας ή άλλου είδους ανικανότητας προς εργασία. Πολύ συχνά λοιπόν δεν γίνεται κατανοητή η οικονομική επίπτωση του να είναι εκτό εργασία το 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στη Σουηδία. Στη Σουηδία αυτό είναι εμφανέ γιατί έχουν καλό σύστημα κοινωνικής ε, ασφάλειας και προστασίας και καταγράφονται όλα αυτά. Είναι όμως ένα γενικευμένο πρόβλημα στο χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα και μεγάλη επιβάρυνση για την κοινωνία. Μαζί με το Φινλανδικό Ινστιτούτο κάναμε κάποιους υπολογισμούς για να υπολογίσουμε την απώλεια από την ανικανότητα προς εργασία πριν από τον χρόνο συνταξιοδότησης. Τα αποτελέσματα από τη Φινλανδία είναι ότι 58,1 είναι η μέση ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ θα περίμενε κανείς 65 έτη και 67 στην Φινλανδία μάλιστα είναι 68 το αναμενόμενο. Αλλά η απώλεια των ε, χρόνων εργασίας είναι 6,9, ε, δηλαδή περίπου 7 έτη από την ενεργό εργασία είναι η απώλεια λόγω της ανικανότητας προς εργασία. Αν ε, εξετάσουμε την απώλεια αυτή είτε σε μία χώρα είτε σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα ότι από την πρόορη συνταξιοδότηση η απώλεια είναι 2,4 ε, δισεκατομμύρια. το 24 πλάσιο των χρημάτων που δώσαμε στην Ελλάδα ή στην Ιρλανδία. Όλα αυτά είναι πόροι που χάνονται λόγω της πρόορης συνταξιοδότησης. Και θα, μπορούσε, θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να εργάζονται περισσότερο αν βελτιώνονταν οι συνθήκες εργασίας. Τέτοια στοιχεία λοιπόν θα έπρεπε να τα λαμβάνουν υπόψη οι Υπουργοί Απασχόλησης. Οι Υπουργοί Απασχόλησης ε, σκέφτονται τα προβλήματα χωρών όπως η Ελλάδα ή η Ιρλανδία, αλλά δεν σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να έχουν τεράστια εξοικονόμηση στην ίδια τους τη χώρα, αν βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να εργάζονται περισσότερο, όχι με διοικητικά μέτρα, αλλά με μέτρα που θα ληφθούν στο χώρο εργασίας, ώστε να είναι ασφαλείς. Εργαζόμενοι ε, που έχουν ε, μειοσκελετικά προβλήματα δεν θα υποφεληθούν από ε, τα μέσα παράτασης του χρόνου εργασίας. Ακόμη και αν η κυβέρνηση παρατείνει τα έτη ενεργού εργασίας, αυτοί που έχουν μειοσκελετικά προβλήματα δεν θα μπορέσουν να εργαστούν περισσότερο. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη οι Υπουργοί Εργασίας. Αν δούμε τώρα τις επενδύσεις, αν δούμε τι επενδύουμε στην αγορά εργασίας, για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, για την καλύτερη ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας και το συγκρίνουμε με τις απώλειες, βλέπουμε ότι οι απώλειες είναι πολύ περισσότερο σημαντικές από τις πραγματικές επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι που προέκυψε από τις εργασίες του δικού μας οργανισμού και θα συνεργαστούμε με τους άλλους οργανισμούς στο μέλλον και ελπίζουμε ότι ε, θα είναι πιο αποτελεσματικά ε, αυτά τα στοιχεία τα οποία θα έχουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Κρίστιαν Λετμάιερ που τελεί χρέη διευθυντού του ΣΕΝΤΕΦΟΠ Η Επιτροπή μας επισκέφθηκε το ΣΕΝΤΕΦΟΠ πέρυσι και καλό θα ήταν να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε σε ό,τι αφορά την έκθεση δραστηριοτήτων, την έκθεση πεπραγμένου και σας παρακαλώ να μην είστε πάρα πολύ μακροσκελείς αν θέλετε να μπορέσετε να απαντήσετε και σε ερωτήματα συναδέλφων μετά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2010 ήταν μια χρονιά όπου το πλαίσιο πολιτικής, το υπόβαθρο πολιτικής ε, ήταν ε, μεταξύ άλλων κατάρτιση και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας μια νέα στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη στον τομέα της κατάρτισης. Εγώ νομίζω ότι, πώς να το πω, Δεν θέλω να φανώ υπερόπτηση ζωνικός, αλλά τα έγγραφα πολιτικής έχουν επηρεαστεί και η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση πλέον έχουν προσλάβει μίζωνα ρόλο για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις σχετικές στρατηγικές. Θα ήθελα να επισημάνω δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας αφενός, μια πρωτοβουλία που βασίζεται σε αποδεκτικά στοιχεία που έχει δώσει το ΣΕΝΤΕΦΟΠ κατά τα προηγούμενα έτη. Ήταν πολύ επιτυχημένη χρόνια του 2010 για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Το Δεκέμβριο παρουσιάσαμε στην Υπουργική Συνάντηση των Υπουργών Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Προύς την έκθεση πεπραγμένων που λάμβανε υπόψη τη δικασία από το 2002 έως το 2010. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν έχει εξελιχθεί, μάλλον δεν έχει ασκήσει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, στην καθημερινή του ζωή, αλλά έχει συμβάλει νομίζω στην πολύ πιο έντονη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των άλλων χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, στη διαδικασία της Κοπενχάγης. Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εργαλείων και των σχετικών αρχών θα αναπτύξει θα αναπτύξει τι πλήρε δυνατότητε όταν υπάρξει εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στη φάση τη εφαρμογή που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη χρονική περίοδο. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων χωρών κάτι πρέπει να παραμείνει. Ένα από τα σημαντικά σκέλη του ΣΕΝΤΕΦΟΠ δεν είναι μόνο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό αυτών των εργαλείων, αυτών των μέσων, αλλά να συνεισφέρει στην φάση της εφαρμογής παρακολουθώντας τις ε, εξελίξεις, την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και βασιζόμενο βέβαια και στην εμπειρία του να προτείνει ενδεχομένω νέες εξελίξεις. Για να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και το ECVET, που είναι το σύστημα μεταφοράς ε, μορίων στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο στόχος μας βέβαια είναι η διαφάνεια και η κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών και έχουμε ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, το Europass, που ευτυχώς βλέπουμε ε, να γίνεται μια από τις σπάνιες περιπτώσεις ε, όπου ένα μέτρο φτάνει στους πολίτες. Ε, πάνω από 17 εκατομμύρια βιογραφικά μεταμορφώνονται, μεταφορτώνονται, συγγνώμη, πολύ πιο πάνω από το στόχο που είχε θέσει ο αρμόδιος επίτροπος Φίγκλ για το 2010. Για να σας δώσω μια ιδέα. Όταν ξεκίνησε το Europass το Φεβρουάριο του 2005, 15.000 μεταφορτώσεις ε, το μήνα έχουν φτάσει στις 300.000 ε, μόνο για τον Οκτώβριο του 2010. Ένα δεύτερο τμήμα των εργασιών μας που ίσως το γνωρίζετε πολύ καλά είναι οι προβλέψεις στον τομέα των αναγκών ε, και της προμήθειας της ε, προσφοράς ε, δεξιοτήτων. Είναι ένα θέμα που η εντολή του ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι να συνεχίσει να επικαιροποιεί τις προβλέψεις αυτές, να τις βελτιώνει, να αναπτύξει περαιτέρω τη μεθοδολογία και αυτό είναι ένα μέρος μόνο της όλης της ιστορίας. Σε ποιο είναι το υπόβαθρο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να έχει σχέση με την αγορά εργασίας. Και αυτό έχει να κάνει και με την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και με τη συνεχή, τη διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Χρειάζεται να διδάξουμε τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας ε, και θα πρέπει να δούμε ποιες αδυναμίες υπάρχουν, οι πράσινε θέσει, παραδείγματος χάρη, ή οι θέσει εργασία που χρειάζονται στον τομέα τη υγεία, λόγω των δημογραφικών συνθήκων. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για τις δεξιότητες και αυτό εντάσσεται στο έργο του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Υπάρχουν επίσης προσπάθειες και συνεισφέρει σε αυτό το έργο και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ για την ανάπτυξη ε, μίας γλώσσας ΕΣΚΟ για τη γεφύρωση των παρανοήσεων μεταξύ κάποιων διατυπώσεων της αγοράς εργασίας, ό,τι αφορά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ανάγκες των, ε, και, και προσόντα τα οποία παρέχει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Βέβαια το ΣΕΝΤΕΦΟΠ συνεχίζει και θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το 2013 να διαχειρίζεται και να συνεισφέρει και στο πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης. 230 επισκέψεις το 2010 οργανώθηκαν με 2.360 συμμετέχοντες. Τώρα ερευνητικό έργο το ΣΕΝΤΕΦΟΠ αξιοποιεί τα ωφέλη της επαγγελματική επένδυσης και κατάρτισης. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί βοηθά να ληφθούν υπόψη επενδυτικέ αποφάσεις των κρατών μελών επενδύσεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το 2011 θα δημοσιευθούν και τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής. Τώρα, της μελέτης. Ό,τι αφορά τα βραχυπρόθεσμα παραδοτέα που φαίνονται και στην ανακοίνωση τη Μπρουζ ίσω υπάρχουν κάποια ζητήματα που κάποιοι θεωρήσουν μια νέα πτυχή των εργασιών του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Θα υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό της ελκυστικότητας ε, της επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτισης. Και θα δούμε και το δίκτυο της κινητικότητας ε, των ε, σπουδαστών. Πιστεύω ε, ότι το Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια μας είχε ζητήσει να αναπτύξουμε μία επικοινωνιακή στρατηγική. Με τα λοιπόν σήμερα να σας ενημερώσω ότι η επικοινωνία, η επικοινωνιακή στρατηγική και η υλοποίησή της ε, υπήρξαν πάρα πολύ επιτυχημένες. Οι ομάδε στόχου και οι βασικοί εμπλεκόμενοι είναι οι χαράκτε πολιτικής βέβαια, αλλά και τα άτομα τα οποία εργάζονται και συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Υπάρχει όμως και ανάγκη να ενημερώσουμε το ευρύτερο κοινό για, την, για τα ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να αναπτύξουμε εργαλεία για να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκομένους φορείς ε, και έχουμε τακτικές δημοσιεύσεις ανακοινοθέντων τύπου για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ επίσης αναβαθμίσαμε και τις προσπάθειές μας για ηλεκτρονική παροχή αυτών των πληροφοριών. Πρόκειται για έργο βέβαια το οποίο θα εξακολουθήσουμε και εντός του 2011 να επιτελούμε Άρα θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες να είναι πιο αποτελεσματικό το ΣΕΝΤΕΦΟΠ με την αυτοματοποίηση των ε, διαδικασιών μας επί παραδείγματι και βέβαια και με την υλοποίηση των συστάσεων των ελεγκτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χουάν Μενέντεθ Βαλντές από το Eurofound, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, με έδρα το Δουβλίνο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, λέγομαι Χουάν Μενέντεθ Βαλντές. Μόλις ε, ανέλαβα καθήκοντα ως διευθυντής από την 1η Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωση και Εργασία στο Δουβλίνο και αποτελεί μεγάλο προνόμιο για μένα να απευθυνθώ σε εσά για πρώτη φορά και να σα παρουσιάσω τα κύρια πορίσματα και τα αποτελέσματα των εργασιών μας για το 2010 αλλά και τα βασικά στοιχεία του επόμενου έτους, του προγράμματος εργασίας για το 2011. Έχουμε το στρατηγικό μας πλαίσιο 2009-2012. Έχουμε στρατηγικούς στόχους για την περίοδο αυτή. Προσπαθούμε να εδραιώσουμε το Eurofound ως μια αξιόπιστη πηγή ποιοτικών πληροφοριών στους τομείς ε, της ε, ειδικότητά μας που είναι οι συνθήκες εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, ε, οι συνθήκες διαβίωσης, ποιότητα ζωής καθώς και η πρόβληψη και διαχείριση των αλλαγών. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τον τριμερή χαρακτήρα και τις σχέσεις μας με τους εμπλεκομένους και να πετύχουμε και την επιχειρησιακή αριστεία. Σε ό,τι αφορά τους στόχους μας, θα ήθελα να σας πω, σε ό,τι το 2010, να σας πω ότι υλοποιήσαμε το 99,5% του προϋπολογισμού που είχαμε στη διάθεσή μας. Άρα παγιώσαμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα του Ιδρύματός μας. Ε, ποια ήταν τα βασικά τώρα ζητήματα στον τομέα της έρευνας. Και αυτό ε, παρά το ότι είχαν οριστεί θεματικές ε, σειρές προτού χτυπήσει το πρόγραμμα εργασίας μας η μεγάλη δημοσιονομική κρίση, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στην κατάσταση και παρουσιάσαμε πορίσματα και σχέδια που είχαν να κάνουν με τον αντίκτυπο της κρίσης ε, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση, την απασχόληση, κοινωνικό διάλογο και την εξέλιξη της εργασίας και της απασχόληση. Επίσης το 2010 κάναμε ένα επιτόπιο έργο και παρουσιάσαμε και τα πρώτα πορίσματα σε μια κοινή εκδήλωση με τη Βελγική Προεδρία σε σχέση με την πέμπτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις ε, συνθήκες εργασίας και βλέπετε ε, ότι έχουμε αποτελέσματα από 34 χώρες με συνεντεύξεις σε 25 γλώσσες και πάνω από 43.000 συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, το Μάρτιο παρουσιάσαμε στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της δεύτερης Ευρωπαϊκής Έρευνας Επιχειρήσεων με στόχο την, με θέματα την ευελιξία και τον κοινωνικό διάλογο. Αλλά είδαμε και άλλους τομείς όπως είναι ο κοινωνικός διάλογος και οι συνθήκες εργασίας, ο αντίκτυπος ε, στις επιδόσεις, επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για τον, τη συμφιλίωση της οικογενικής και της εργασιακής ζωής και επίσης τα θέματα της αλληλεγγύης για μετανάστες, νεαρά άτομα με αναπηρία ή προβλήματα υγείας. Είχαμε σημαντικές ασκήσεις συλλογή δεδομένων και ανάλυσης ε, μέσω των ευρωπαϊκών ερευνών αλλά και των παρατηρητηρίων μας των τριών παρατηρητηρίων. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Προσπαθήσαμε τις τελευταίες χρονιές και θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε και στο μέλλον τη συνεργασία μας με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και θα προσπαθήσουμε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των δραστηριοτήτων μας. Άρα θα έχουμε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους διάφορους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και τη στενή συνεργασία με αδελφούς οργανισμούς υπάρχουν ε, διαφορετικές συμφωνίες και μνημόνια συνεννόησης. Επίσης, συνεργαζόμαστε και με άλλους διεθνούς οργανισμούς σε διάφορα project, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Εργασίας και ο ΩΣΑ. Τώρα έρχομαι στο πρόγραμμα εργασίας για το 2011. Είναι σταθερός ο προπολογισμό μας, ε, ανέρχεται σε 20 περίπου εκατομμύρια ευρώ Βλέπετε στις διαφάνειες τι δραστηριότητές μας και το μερίδιο του προπλησμού που αντιστοιχεί. Βλέπετε ότι στις κύριες δραστηριότητες του Ιδρύματος είναι το 80% των πόρων. Δηλαδή παρατηρητήρια, έρευνες, απασχόληση ανταγωνιστικότητα, εργασιακέ σχέσεις, συνθήκες διαβίωσης, πληροφορία, πληροφορήση και ενημέρωση. Το 2011 θα συνεχίσουμε επίσης ε, και κάποια έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά θα αναπτύξουμε και νέα έργα στους τρεις βασικούς τομείς έρευνας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη απασχόληση στις μεταλλασσόμενες αγορές εργασίας έχουμε το θέμα flexicurity ευελιξία με ασφάλεια την αναδιάρθρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, την πρόβλεψη και διαχείριση της επίπτωσης του πρασινίσματος ε, των βιομηχανιών και απασχόληση νέων, ιδίως προκλήσεις και λύσεις για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας. Επίση, άλλο άξονα, περισσότερε και καλύτερε θέσει εργασία. Θα ξεκινήσουμε έργα σε ό,τι αφορά εθνικέ πρακτικέ για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων με βάση τον κανονισμό των εφιστάμενων. Θα δούμε επίση την οργάνωση εργασία, την καινοτομία και τι συνθήκε εργασία και εργασιακέ σχέσει στον δημόσιο τομέα. Τρίτο άξονα προώθηση τη κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη κοινωνική προστασία. Θα έχουμε κάποια σχέδια κινητικότητα και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Θα δούμε επίσης τις συνθήκες ε, διαβίωσης των Ρωμά καθώς και το εισόδημα μετά τη σύνταξη. Σε ό,τι αφορά τις έρευνες, θα έχουμε το επιτόπιο έργο κατά το 2011 για την τρίτη Ευρωπαϊκή Έρευνα Ποιότητας Ζωής. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε το ερωτηματολόγιο και μετά θα ξεκινήσει το επιτόπιο έργο. Θα αναλύσουμε επίσης στοιχεία που έχουμε από το Ευρωβαρόμετρο από τις χρονιές 2009 και 2010 πάντα για τις συνθήκες διαβίωσης και επίσης θα κάνουμε μια ανασκόπηση και θα εκπονήσουμε εκθέσεις από τη δευτερογενή ανάλυση των δεδομένων από την πέμπτη Ευρωπαϊκή Έρευνα ε, Συνθήκων Εργασίας που την ανέφερα πριν με εστίαση στην ευελιξία του ωραρίου εργασίας, την ισορροπία ιδιωτικού βίου και επαγγελματικού βίου, ποιότητα εργασίας και απασχόλησης, απασχολησιμότητα και ασφάλεια και επίσης θα κάνουμε και μια νέα δευτερογενή ανάλυση των δεδομένων δεδομένων της δεύτερης ευρωπαϊκής ε, έρευνας για τις επιχειρήσεις. Επίσης, τα τρία παρατηρητήριά μας ε, θα συνεχίσουν να εργάζονται, θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε επικαιροποιημένα δεδομένα, να τονίσω κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τις ε, επικαιροποιήσεις, τις επικαιροποιήσεις για την αμοιβή, για την, το χρόνο εργασίας, Είχαμε επίσης κάποιες εκθέσεις ε, για την ε, ΔΕΛΤΑΓΑΜΑ απασχόληση και την ετήσια έκθεση του ERM. Επίσης θα παρουσιάσουμε 10 συγκριτικές αναλυτικές εκθέσεις βάσει των εθνικών εκθέσεων ε, των κρατών μελών. Θα σας αναφέρω τρία, τρία θέματα. Βλέπετε στη διαφάνεια η εξέλιξη των μισθών στη διάρκεια της κρίσης, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές για, τους, για τα επιδόματα ανεργίας και οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής σε σχέση με την με την απασχόληση των νέων και επίση θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τομεακέ συγκριτικέ εκθέσει και μελέτες αντιπροσωπευτικότητα. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τομεακού Διαλόγου. Επόμενη διαφάνεια. Θα θέλαμε επίσης και σε εσωτερικό επίπεδο να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις δικές μας επιδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε το σύστημα μέτρησης ε, των επιδόσεών μας, όπου θα μετρούμε ζητήματα όπως είναι ο αριθμός των χρηστών ε, ή των μεταφορτώσεων εγγράφων από τις ιστοσελίδες μας, ε, κάποια έγγραφα πολιτικής, παρουσιάσεις, επαφές με χαράκτες πολιτικής Θα πρέπει επίσης να υλοποιήσουμε και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τα διάφορα σχέδια γράσης μετά τις συστάσεις ε, της εσωτερικής υπηρεσίας ε, ελεγκτών. Έχουμε το 2011 έλεγχο της ε, διαδικασίας διαχείρισης των ερευνών του Eurofound θα προχωρήσουμε επίσης και στην εξ αξιολόγηση του πρόγραμματος εργασία για τα 2005-2008 και κάποια άλλα πιο εξειδικευμένα θέματα. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να τονίσω το εξή: Πέραν τη υλοποίηση του προγράμματο εργασία μας για το 2011, Μία από τι προκλήσει που έχω να αντιμετωπίσω είναι να ε, δω προ το μέλλον και να προσπαθήσω ήδη ε, ευθύ εξ αρχή να προετοιμάσω το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2012 καθώς και ένα νέο πλαίσιο ε, για, το επόμενο, για την επόμενη τετραετία. Εμείς ε, διατηρούμε σταθερά τις επαφές με τους ε, διάφορους ενδιαφερομένους φορείς με τους συντονιστές και τους ηγητές από πλευράς Κοινοβουλίου έχουμε συχνές επαφές και φυσικά θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον οποιασδήποτε συστάσεις έχετε να διατυπώσετε. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε στα πλαίσια ε, της παρουσίασής σας για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας και βεβαίως σας ευχόμαστε ε, ό,τι καλύτερο ε, στην εργασία σας. Τελευταία, αλλά όχι ελάσσονος σημασίας, είναι η τελευταία μας παρουσίαση λοιπόν της ΕΤΕΦ με έδρα στο Τωρίνο και είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ε, τον οργανισμό του οποίου επικεφαλής είναι η κυρία Σερβάνα ε, στην αρχή του χρόνου. Ε, θα ήθελα πριν σας δώσω το λόγο κυρία Σερβάνα να σημειώσω ότι βρίσκονται μεταξύ ημών οι δύο εμπειρογνώμονες που όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού ε, ETF, ο κύριος Φρανσουά Μεζιέρ και η κυρία Σάρα Πάρκιν οργάνωσαν ε, ένα side meeting, μια παράπλευρη οργάνωση, ε, συνάντηση, ε, κατά την οποία μετά τις 6.30 θα μπορέσετε να ανταλλάξετε απόψεις. Κύριε Σερμπάν, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα πρώτα απ' όλα να, ευχαρισ... σας ευχηθώ ευτυχές το νέο έτος 2011. Ε, και τα καλύτερα σε εσά αλλά και τους πολίτες της Ευρώπης. Έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου και πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, το ETF, είναι το μόνο το οποίο συνεργάζεται και με συνδεδεμένες ε, χώρες, εκτός δηλαδή των ε, χωρών που είναι πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουλεύουμε σε 29 χώρες και το τονίζω, γιατί στα τέλη του 2010 ξεκινήσαμε συνεργασία και με την Ισλανδία και επομένως ε, για το 2011 πλέον μιλάμε για συνεργασία με 30 και δραστηριότητες σε 30 ε, χώρες ε, μέλη. Εργαζόμαστε με τις χώρες αυτές έτσι ώστε να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν ένα καλό σύστημα κατάρτισης το οποίο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και θα οδηγήσει σε την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Επίσης προσπαθούμε να συμβάλλουμε ε, στην ε, ε, συνολική εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσουμε σε συνεργασία με τις χώρες αυτές να τις βοηθήσουμε να διαμορφώσουν καλύτερα την παγκοσμιοποίηση και να εκμεταλλευτούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες ε, υπάρχουν κάποιες ε, θεματικές ε, προσεγγίσεις τις οποίες εγκρίνεται το 2008 και πλέον είχαμε το δεύτερο έτος εφαρμογής από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης της αναδιατυπωμένης οδηγίας το 2010 εστιάσαμε την προσοχή μας στις ολοκληρωμένες πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση οι χώρες να εφαρμόσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ε, καλής ποιότητος προγράμματα ε, κατάρτισης που θα μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην οικονομική και λοιπή ανάπτυξη και που θα οδηγήσουν τελικά σε λιγότερη φτώχεια και λιγότερες, λιγότερες στερήσεις γιατί υπάρχουν ε, κάποια προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ αναπτυγμένα και χώρες ε, οι οποίες έχουν προχωρήσει ε, πάρα πολύ όπως η Κροατία ας πούμε ή όπως η Ισλανδία αλλά έχουμε και χώρες όπου η φτώχεια είναι μια κατάσταση καθημερινή και προσπαθούν και αγωνίζονται να επιβιώσουν μέρα με την ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι οι δραστηριότητες μας όλες έχουν τεθεί υπό, την, ε, ε, υπό το γενικότερο πλαίσιο του έτους 2010 που ήταν ε, το έτος καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά αυτή την έννοια οργανώσαμε κυρίως για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έναν διάλογο βάσει συγκεκριμένων πολιτικών θεμάτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε ε, τα στοιχεία τα οποία μπορούν καλύτερα να οδηγήσουν σε ανάπτυξη τα Δυτικά Βαλκάνια και πρέπει να πω ότι δουλεύουμε ε, βοηθώντας τις χώρες βεβαίως αλλά και προωθώντας ε, την περιφερειακή συνεργασία των χωρών αυτών πράγμα όχι πάντα πολύ εύκολο. Όμως είναι βέβαιο και σας το λέμε εδώ η επαγγελματική ε, κατάρτιση ε, και ε, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό συνεργασίας και ανάπτυξης. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να υπογραμμίσω το γεγονός ότι εργαζόμαστε βάσει ανάλυσης πολιτικής, στηρίζουμε τον, την πολιτική διαλόγου, την πολιτική ανάπτυξης, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας πούμε, πηγαίνοντας, όπως είπα και προηγουμένως, στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και εκεί, ε, σαν αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μας, ε, έχουμε καταφέρει να λύσουμε εν μέρη το πρόβλημα των χωρών αυτών όσον αφορά ε, τον κοινωνικό αποκλεισμό, ας πούμε, όσον αφορά την κοινωνική περιθεριοποίηση, γιατί υπάρχουν εκεί ε, πολίτες στους οποίους ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες έτσι ώστε να τους βοηθήσουν με τη σειρά τους ε, θέλει η επιτροπή να βοηθήσουμε τις χώρες της νοτιοανατολικής ευρώπης έτσι ώστε να αναπτυχθεί και ο ιδιωτικός τους τομέας. πώς είναι δυνατόν όμως να πετύχουμε κάτι τέτοιο χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες. γι' αυτό λοιπόν εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην συνεργασία με τις χώρες έτσι ώστε και από πλευρά των χωρών να υπάρχουν οι δεξιότητες τις οποίες ζητούμε και τις οποίες η ίδια η κοινωνία ζητάει οι ίδιες οι χώρες θα πρέπει να εξεύρουν αυτές τις μακρό, μακρόπνοες και μακρόχρονες πολιτικές οι οποίες θα τους βοηθήσουν, θα βοηθήσουν τις ίδιες τις χώρες πρώτα απ' όλα. Επίσης, εμείς ελπίζομαι ότι Ήδη μέσα στο 2011 θα έχουμε την δυνατότητα ε, να έχουμε την πρώτη έκθεση των πεπραγμένων των χωρών αυτών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να έρθετε 10 και 11 Μαΐου στο Τωρίνο για να ακούσετε κι εσείς αυτές τις εκθέσεις πεπραγμένων. Ε, εμείς δουλεύουμε πολύ με όλα τα θεσμικά όργανα των κοινωνικών εταίρων έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα διαλόγου μεταξύ αυτών των οργανισμών και των κυβερνήσεων με ε, κύριο επιζητούμενο το, την επίλυση προβλημάτων κυρίως στην νότια μεσογειακή ε, περιοχή ε, η δυνατότητα ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων ε, μπορεί να μας οδηγήσει στην εξέβρεση των σωστών δεξιοτήτων αλλά και στην δημιουργία των ευκαιριών κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία των δεξιοτήτων που χρειάζεται η χώρα. Επίσης, ε, εργαζόμαστε βάσει του σχεδίου που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές. Και αναφέρομαι εδώ σε χώρες οι οποίες είναι ήδη, ε, ήδη σε διαδικασία ένταξης, αλλά και αυτές οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να ε, ενταχθούν. Η με την Μολδαβία, με την Γεωργία και το 2011 θα ξεκινήσουμε με την Αρμενία το λεγόμενο Mobility Partnership. Τι είναι αυτό. Ε, είναι η ε, προσπάθεια στήριξης της επιστροφής μεταναστών από την Ευρώπη στις χώρες τους. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ε, έχει κανείς την απαραίτητη εμπειρία και την αναγνώριση των των ε, δεξιοτήτων του. Και εδώ ε, θα συμφωνήσω με τα όσα ο πρόεδρος Σεντεφόπ είπε προηγουμένως ε, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών κτλ. Βοηθούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και μέσω της εταιρικής σχέσης κινητικότητας, mobility partnership, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους αναγνώρισης της εμπειρίας και των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Αυτή είναι η εξωτερική διάσταση των πλαισίων ε, προσόντων ε, που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα, αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα αναγνώρισης ικανοτήτων και δεξιοτήτων και προσόντων και πρέπει να σας πω, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ότι τον, ε, τον Οκτώβριο υπό Πολωνική Προεδρία θα ξεκινήσουμε ένα ε, διάλογο και ένα πρόγραμμα ε, στα πλαίσια του οποίου θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω εικονικής πραγματικότητας να δουν όλα τα μέλη του τι γίνεται στην Ευρώπη. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που ήρθα σήμερα εδώ και χαίρομαι που μπόρεσα να σας πω όλα αυτά που κάνει κάνει το ε, Ίδρυμά μας. Και στα λίγα λεπτά που μου μένουν να σας πω ότι το 2011 υπό Ουγγρική Προεδρία θα ξεκινήσουμε την εργασία για το πλαίσιο ε, προσόντων ε, μέσω ολοκληρωμένης στρατηγικής. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά ε, κράτη-μέλη και μη κράτη-μέλη έτσι ώστε να συνδυαστούν, να δουλέψουν μαζί, να δουν πώς είναι δυνατόν η καινοτομία, τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν σε πολυετή βάση να βοηθήσουν τις χώρες αυτές. Και επίσης συνεχίζουμε την εργασία με ε, το, την Επιτροπή ε, των, με την Επιτροπή των Περιφερειών ε, για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Ο γείτονά μου αναφέρθηκε προηγουμένω στι ε, δεσμεύσει και πρέπει να σα πω ότι ε, για το δεύτερο μισό του ε, μέρου, του έτου, συγγνώμη, έχουμε από άποψη δημοσιονομική καλυμμένο το 99,9% του προϋπολογισμού μας και αυτό μετά την αδιατύπωση της οδηγίας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Όσον αφορά τώρα ε, το 2011 ε, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν οι δημοσιονομικές προοπτικές για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης στα πλαίσια της στρατηγικής 20. And uh, therefore we will be extremely if in 2011... Ε, θα ήμουν ε, απολύτως ευτυχής εάν ε, το 2011 θα μπορούσατε να μας επισκεφτείτε για να δείτε από κοντά τι κάνουμε σε όλες τις χώρες. Συγγνώμη, αλλά έχασα τη φωνή μου, όχι όμως και τη ρόμη της παρέμβασής μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάω στους εγγεγραμμένους ομιλητές, αλλά πριν τους δώσω το λόγο, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπουλόν, που έρχεται μετά την αποχώρηση της κυρίας Πασκάλ Μπρουνί και θα ήθελα να τον καλωσορίσω εκ μέρους όλων μας και ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα είναι εξίσου επικοδομητική όπως είχαμε και με την κυρία Μπρουνί ε, που πέρασε στην Εθνική Βουλή. Πριν σας δώσω το λόγο όμως θα ήθελα και εγώ ίδια να κάνω δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Γιούγκα Τάκαλα καταρχήν για τη μελέτη ε, την οποία ε, ε, εσείς ξεκινήσατε, την SNR. Τι διδάγματα μπορούμε εμείς ως νομοθετικό όργανο να εξαγάγουμε όσον αφορά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύετε ότι για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους υπάρχουν κάποιοι τομείς και σας ζητάω εδώ να βγείτε λίγο από το ρόλο ε, του διενεργήσαντος τη μελέτη και να μας ε, πείτε ε, από την οπτική γωνία της πρακτικής εφαρμογής τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πού θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση με βάση τα στοιχεία της μελέτης την οποία διεξαγάγατε και προς την κυρία Σαρμπάν. Ξέρω ότι εσείς εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά με βάση τα όσα έγιναν στην Τινησία που ίσως κάπως να είχαν ε, υποπέσει στην αντίληψη του Ιδρύματος ε, ως πρόβλεψη. Τι διδάγματα ε, μπορείτε να συναγάγετε. Ιδίως όσον αφορά την πλαισίωση προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας, ιδίως σε τομείς όπως είναι ο δικαστικός τομέας και η κατάρτιση των δικαστών, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα οι μηχανισμοί και να εκλείψουν οι μηχανισμοί διαφθοράς. Θα αναθεωρήσετε κάπως τον προγραμματισμό σας, το είχατε ήδη προβλέψει, αλλά ακόμη και αν είχατε προβλέψει κάτι, νομίζω ότι με τις εξελίξεις στην Τινησία υπάρχουν σίγουρα αλλαγές. Επανεξετάζετε τον προγραμματισμό σας με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή μας για τη συζήτηση και έχουν ζητήσει το λόγο τουλάχιστον 7 συνάδελφοι. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να είστε όλοι πολύ σύντομοι. Ο κύριος Σαρκάς και μετά η κυρία Μογά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Γιατί θα αναφερθούν σε κάποιους συγκεκριμένους οργανισμούς άλλοι σοσιαλιστές συνάδελφοι. Θα ήθελα στους ε, τρεις διευθυντές και τη μία διευθύντρια να τους καλωσορίσω όλους εξ ονόματος ε, των σοσιαλιστών βουλευτών να τους επαναλάβω και την αναγνώρισή μας προς το έργο το οποίο επιτελούν για την ορθή εφαρμογή των πολιτικών που άπτονται του δικού μας πεδίου αρμοδιοτήτων. Θέλω να πω ότι στη δική μας ομάδα εργασίας αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι όχι μόνο να παρακολουθούμε την εξέλιξη στην αγορά εργασίας και την τρέχουσα κατάσταση, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε κάποιες ε, εκτιμήσεις, προβλέψεις, να προεξοφλήσουμε ίσως κάτι το οποίο ε, προαναγγέλλεται, δηλαδή αλλαγή, μια νέα μέθοδο παραγωγής, νέα μέθοδο εργασίας. Και όλα αυτά ε, πιστεύω ότι απαιτούν από τις τέσσερις συνιστώσεις, δηλαδή από τους τέσσερις οργανισμούς και την ικανότητα πρόβλεψης, πρόγνωσης αν θέλετε του μέλλοντος, αλλά και προσαρμογή στην πραγματικότητα. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Ούτε σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ούτε σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, σε κανέναν από του τομεί που για τους οποίους εργάζεστε και εσείς και εμείς. Τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ όπως πριν. Και είναι πραγματικά πολύτιμη δουλειά που επιτελείτε στους οργανισμούς σας και θέλω να σας εμψυχώσω, και να σας πω ότι πρέπει να συνεχίσετε αυτή την άσκηση πρόβλεψης. Τώρα, στον κύριο Λεν το λέω κάθε χρόνο σχεδόν, ε, η ανησυχία μου δεν πρέπει να παραμένουν κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα κρατάμε μέσα μας, αλλά πρέπει να τα βγάζουμε προς τα έξω. Και θα πρέπει να δούμε και με τις επιχειρήσεις, με την κοινότητα των πολιτών, με τους ε, πολίτες, με τα συνδικάτα, ε, να τους διαδώσουμε, να τους ενημερώσουμε και όχι μόνο να συνεχιστούν οι πολιτικές αυτές επικοινωνίας που έχετε, αλλά και να αυξηθούν, να διευρυνθούν. Και αν μου επιτρέπετε μία παρατήρηση να καλωσορίσω και εγώ ε, τον ε, Διευθυντή Eurofound και συμπατριώτη μου, τον κύριο Μενέντεθ Βαλντές. Και να σας πω κύριε Βαλντές, ε, οι άλλοι το γνωρίζουν, αλλά αφού μόλι αναλάβετε τα καθήκοντά σας, πρέπει να σας πω ότι εδώ θα έχετε μόνο φίλους. Είναι σκληρή η κοινοβουλευτική ζωή και οι βουλευτές πάντοτε είναι αυστηροί με τις κυβερνήσεις. εδώ πρέπει να σας πω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Είμαστε φίλοι σας, θα συνεργαστούμε χέρι με χέρι. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. κυρία Μοχά και μετά η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους τέσσερις ε, διευθύντες των οργανισμών που έλαβαν ε, το λόγο και έκαναν τις παρουσιάσεις τους. Πριν συνεργαστούμε με αυτούς τους οργανισμούς ε, ήμουν κάπως διστακτική γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός οργανισμών αλλά ε, όταν σας επισκέφθηκα επί τόπου, όταν ε, άκουσα αυτά που είχατε να μας πείτε και βλέποντας τις μελέτες τις οποίες παράγετε, σήμερα μπορώ να σας πω ότι είμαι βεβαία για ένα πράγμα ότι δεν εκμεταλλευόμαθα πλήρως τις εργασίες ε, τις δικές σας γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι δραστηριότητές σας και μπορούν να μας διαφωτίσουν σε πολλές πτυχές των δραστηριοτήτων μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την ε, πολύ σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας που κάνατε. Έχω άλλες ε, δύο ερωτήσεις ε, προς τον Διευθυντή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Πρώτον, είπατε ότι το 1 τρίτο των εργαζομένων απουσιάζουν από το χώρο εργασίας τους. Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε αυτό. Γιατί απουσιάζουν και τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να καταλογίσουμε καλύτερα ε, την απώλεια χρόνου εργασίας από την πρόορη συνταξιοδότηση. βλέπουμε τα πολύ ψηλά χρηματικά ποσά τα οποία χάνονται ακριβώς λόγω της πρόορης αποχώρησης των εργαζομένων και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις πατάλες. Επίσης έχω μια ερώτηση προς το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Θέλω να επαναλάβω εδώ ενώπιόν σας πρόεδρε πόσο η αποστολή την οποία κάναμε στο Σεντεφόπ τον Νοέμβριο, τότε που εσείς είχατε πάει στο Τωρίνο Πρόεδρε, είχαμε πάει εμείς στο Σεντεφόπ, με την Άντια και την κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψή μας. Ιδίως για το θέμα των νέων προσόντων για τις νέες θέσεις απασχόλησης Αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε πολλά για, για την εξέλιξη της εργασίας και για το Europass και για το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα. Αυτά τα οποία πληροφορηθήκαμε ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν ε, να έχουμε νέες δεξιότητες για τις νέες θέσεις απασχόλησης και για μας είναι δύσκολο πρόβλημα το να εξασφαλίσουμε την εξέλιξη αυτών που ήδη βρίσκονται στην αγορά εργασίας προς τις νέες δεξιότητες. Τι συμβουλές θα μπορούσατε να μας δώσετε εσείς και ποιες είναι οι απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές. Προς την κυρία Σερμπάν, τέλος θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών διότι δεν ε, δουλεύουν απομονωμένα αλλά συνεργάζονται και επίσης είναι σημαντικό να υπάρχουν περιφερειακές στρατηγικές μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και γειτονικών χωρών όπως είναι η στρατηγική στην περιοχή του Δούναβη, κάτι το οποίο σίγουρα θα είναι προς όφελος των μελλοντικών εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η κυρία Γενιά και η κυρία Χίρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εκπροσωπησή σας εδώ και θα ήθελα ιδίως ε, να απευθυνθώ στον ε, Διευθυντή του Οργανισμού του Δουβλίνου. Ε, με ενδιαφέρον πάρα πολύ αυτό το οποίο είπατε για την απασχόληση και την απασχόληση των νέων και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Επίσης θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι ε, για μας ότι ε, σε ε, περιόδους κρίσης κάνετε τις μελέτες αυτές γιατί η δουλειά σας είναι πολύ σημαντική ιδίως σε περίοδους κρίσης για να έχουμε μελέτες και αποτελέσματα επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ακόμη θέλω να τονίσω ότι θεωρώ πολύ σημαντική τη συνεργασία την οποία είχατε με άλλους φορείς όπως είναι ο ΣΑ ή το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η εντατικοποίηση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς σίγουρα θα προσφέρει ε, πολλά και πολλές πληροφορίες. Θεωρώ πολύ σημαντικές τις δραστηριότητές σας και χαιρετίζω κάθε εντατικοποίηση της συνεργασίας ε, και για την εξέλιξη του κλίματος εργασίας, ε, για τη διαμόρφωση δικτών για την εργασία και επιθυμούμε να εντατικοποιηθεί η, εργασία, η συνεργασία στο μέλλον. Κυρία Χίευς και κυρία Στάινοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν και εκ μέρους των φιλελευθέρων θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους διευθυντές των οργανισμών που μας έκαναν τις παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων τους. Είπαν πολλά οι προηγούμενοι ομιλητές και δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω απλώς και να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό για μας και για μένα συγκεκριμένα που είμαι ε, ε, ε, νέα βουλευτής. Ήταν πολύ χρήσιμες οι επισκέψεις που κάναμε. Το Νοέμβριο συμμετείχα και εγώ σε αυτήν την επίσκεψη. Ήταν χρήσιμο να δούμε την εξειδίκευση και τις νέες πληροφορίες. Εγώ είμαι εισηγήτρια για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και θέλω να τονίσω ότι με βοήθησε πάρα πολύ επιτόπου επίσκεψη γιατί μας δόθηκαν και οι κατάλληλες πηγές και οι μελέτες οι οποίες γίνονται και οι επαφές ε, τις οποίες μπορούμε να έχουμε. Πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για μας ε, τους ευρωβουλευτές, γιατί ξέρει ο καθένας ε, την δική του χώρα, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλος πλούτος πληροφοριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τις πηγές που μας αποκαλύψατε και για την πολύ καλή συνεργασία και περιμένω και τη μελλοντική μα συνεργασία με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Κυρία και κύριο Στερόσα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλους ε, και ιδίως προς την Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Είδα το πρόγραμμα εργασιών σας για το 2011 και άκουσα και τις παρουσιάσεις, τις παρουσιάσεις για το παρελθόν. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να μπορούμε να εξάγουμε τα προγράμματα κατάρτισης και την εμπειρία μας και στις ε, τρίτες χώρες. Ε, ήμασταν προσφάτως στο Κωσυφοπαίδιο και μιλήσαμε με εκπροσώπους οργανώσεων νέων ε, και επαγγελματικής κατάρτισης και είδαμε ότι είναι μεγάλη η ανάγκη για καλή εκπαίδευση και κατάρτιση. Αποτελεί και προϋπόθεση για σωστή αγορά εργασίας για να μην υπάρξει μια αρνητική επίπτωση, αντιθέτως να υπάρξουν μόνο θετικές επιπτώσεις. Για τις χώρες εταίρους θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ποιες είναι οι σημαντικές χώρες εταίροι. Είπατε επίσης ότι από τις χώρες εταίρους παίρνετε κάποια θέματα. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα σημαντικά θέματα για τις χώρες εταίρους και ποια είναι τα δικά σας σημαντικά θέματα για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προίνσης Ντερόσα και η κυρία Edith Bauer μετά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οργανισμούς. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για τον Οργανισμό για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Όπως ε, αναφέρεται στην Ελληνία τις τελευταίες εβδομάδες, ο αριθμός των θανάτων στη Γεωργία έχει διπλασιαστεί. Νομίζω κατά το προηγούμενο σε σχέση με το πρώτο προηγούμενο. Και υπάρχει μια τάση προς τα κάτω, μια πτωτική τάση. Κάτι τέτοιο ε, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια έρευνα, διερεύνηση του αιτίου. Είναι συμπτωματικό. Υποδηλώνει αποτυχία συστημάτων, αστοχία συστημάτων. Τι ακριβώς ε, ε συμβαίνει αυτό. Είναι μια τάση στην Ευρώπη. Στη Γεωργία, ιδίως στην Ιρλανδία, Φαντάζομαι ότι πολλοί εργάζονται ατομικά με μηχανήματα και ζώα και ίσως υπάρχουν σίγουρα κίνδυνοι ε, αυξημένοι για κάποιο ατύχημα. Τώρα, να καλωσορίσω τον νέο διευθυντή του Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας και αφού είναι στην πατρίδα μου το Δουβλίνο, ελπίζω σύντομα να μπορέσω να το επισκεφθώ. Το ερώτημά μου αφορά την έννοια ευελιξία με ασφάλεια, flexicurity. Είπατε ότι εκπονήσατε μια έκθεση για την ευελιξία και ασφάλεια εντό των επιχειρήσεων κτλ. και θα ξεκινήσετε μια έρευνα για τις πρακτικές flexicurity στις επιχειρήσεις. Με εκπλήσει το γεγονό ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια τουλάχιστον υπάρχει μια τάση προ την ευελιξία αλλά με λιγότερη ασφάλεια. Δηλαδή όλο και μεγαλύτερη είναι η ανασφάλεια στο χώρο εργασίας λόγω και της ε, κρίσης ε, που σοβεί σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που το εξετάζεται και θα το εξετάσετε και στο πλαίσιο της νέας μελέτης που θα εκπονήσετε. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποια είναι, ε, ποιος, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη μελέτη αυτή και τι πεδίο εφαρμογή θα έχει. Θα καλύψει κάποια συγκεκριμένα ή όλα τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο ερώτημά μου έχει να κάνει με το νέο έργο που προβλέπεται, ένα νέο σχέδιο για έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο. Μιλάμε για το δημόσιο τομέα ή για κρατικές επιχειρήσεις για τους δημόσιους λειτουργούς ή γενικότερα για τις ε, δημόσιες επιχειρήσεις. Και ένα τελευταίο ερώτημα και συγγνώμη που έχω κάνει τόσες πολλές ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τι συνθήκε διαβίωση των Ρωμά. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Διερωτώ με αν αυτό θα καλύπτει κάτι που είναι ένα πρόβλημα τουλάχιστον στην Ιρλανδία για τους πλανόδιους αν Δηλαδή αντιμετωπίζετε διαφορετικά τις δύο αυτές κατηγορίες ή με τον ίδιο τρόπο. Γιατί σίγουρα οι πλανόδοι ταξιδιώτες υπερβαίνουν κατά πολύ τους Ρωμά. Αλλά δεν είναι και καλύτερες οι συνθήκες διαβίωσής τους. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προτίθεστε ακριβώς να μελετήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντε Ρώσα, θα πάμε στο Δουβλίνο 20 και 21 Ιουνίου. Για να το σημειώσετε, σας το λέω αυτό. Εκτός αν δεν υπάρξει πρόβλημα. Και 17-18 Μαΐου θα πάμε στο Μπιλμπάου. Οπότε, όπως ήθιστε, θα καλύψουμε όλους τους οργανισμούς μέσα στη διετία. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους εκπροσώπους των οργανισμών ε, για το σεβασμό που τρέφουμε στο πρόσωπό τους. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Για την Επιτροπή μας είναι πραγματικά αναγκαίοι όλοι οι οργανισμοί. Θα ήθελα να προσθέσω δύο ερωτήματα σε αυτά που έχουν ήδη τεθεί. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο Τάκουλα. Έχετε στοιχεία, θα ήθελα να γνωρίζω, σε σχέση με την πρόορη συνταξιοδότηση και σε ποιο βαθμό αυτή αφορά γυναίκες και άνδρες. Έχετε κάποια πιο αναλυτικά στοιχεία. Και γιατί, αν υπάρχει, υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Σεντεφόπ το εξή. Αν θυμάμαι καλά, είχατε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την είχαμε δει και εδώ στην Επιτροπή μας σε σχέση με 19 τομείς της οικονομίας, αν δεν απατώμε. Παρουσιάζονται τα στοιχεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και κάποια προκαταρκτικά δεδομένα. Και σε ό,τι αφορά τα πορίσματα της έρευνας σας, είχατε επισημάνει ότι είναι πολύ σημαντικά τα προσόντα για το μέλλον λόγω των αλλαγών, λόγω της κινητικότητας ε, που χαρακτηρίζει την οικονομία. Πότε όμως θα έχουμε τα οριστικά πορίσματα της μελέτης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις όλους τους ε, εκπροσώπους των οργανισμών. Και θα ήθελα να μιλήσω για την εξέλιξη της εργασίας τα τελευταία 30 χρόνια. Ξέρω ότι σήμερα κινούμεθα προς μια εντατικοποίηση της εργασίας. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων μέσα στις επιχειρήσεις ε, και δημιουργείται ένα δυσάρεστο κλίμα μέσα στις επιχειρήσεις υπενθυμίσατε εσείς τις διαταραχές τις μυοσκελετικές καθώς ε, και την ε, αύξηση των ψυχοκοινωνικών ε, κινδύνων. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και ανακαλύπτουμε ότι η εργασία σκοτώνει λόγω των ατυχημάτων, λόγω των επαγγελματικών ασθενειών και λόγω προσωπικών επίσης παραγόντων. Η ερώτησή μου είναι τι πολιτικές πρόληψης υπάρχουν τι ρόλο αποδίδεται στην ε, ιατρική στους χώρους εργασίας. Τι κάνετε για να ε, ακούτε τις προειδοποιήσεις που προέρχονται από τους εργαζομένους. Γιατί οι εργαζόμενοι που καμιά φορά κρούν τον, κίνδυνα, τον κόδωνα του κινδύνου, αντί να εισακουστούν, ε, παραμερίζονται και μπαίνουν στο ψυγείο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προλαμβάνουμε τα προβλήματα. Οι συνθήκες εργασίας σήμερα με την γενίκευση του μοντέλου εργασίας που έχουμε προϋποθέτει κινδύνους όπως είναι κίνδυνοι από χημικά προϊόντα από τα οποία κινδυνεύουν οι έγκυοι γυναίκες που μετά από λίγα χρόνια ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν από διάφορες μορφές καρκίνου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, πολύ. Πρόεδρος. Ελπίζω οι τέσσερις διευθυντές των οργανισμών να σημείωσαν όλες τις ερωτήσεις. Ακούγοντα κανεί όλε τι ερωτήσει, έχει την εντύπωση ότι ήμασταν σε ένα πολυκατάστημα όπου από κάθε ράφι είχαμε και κάτι να πάρουμε. Άρα έχετε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων στι οποίε πρέπει να απαντήσετε και σας παρακαλώ να επικεντρώσετε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στο δικό σας οργανισμό ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε με αντίστροφη σειρά και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σερμπάν καταρχήν για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να πω, να επικεντρωθώ στην κατάσταση στην Τινησία. Ήδη την προηγούμενη χρονιά το Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ε, είχε αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτών των χωρών και προσπάθησε να μάθει από τα μαθήματα των περιοχών. Στις εξωτερικές σχέσεις ε, ε, όταν βασιζόμαστε στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ε, και τις επαγγελματικέ καταρτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερόμαστε στο ε, ευρωπαϊκό κεκτημένο και την, τον κοινωνικό διάλογο που αποτελεί ένα από τα κυριότερα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου. Άρα να μην εργαζόμαστε μονάχα με τις κυβερνήσεις αλλά και με όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς στις χώρες. Επομένως έτσι ο διάλογος με τις αντίστοιχε χώρες ε, παίρνει μια νέα όθηση. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι εμείς τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε σε επίπεδο στρατηγικής. Ε, όταν ε, ε, είναι συμμεριζόμενες, είναι μοιρασμένες οι αρχές αυτής της στρατηγικής, τότε είναι λίγο πιο εύκολο να δουλέψει κανείς. Επίσης μειώνεται το φαινόμενο της διαφθορά, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ελέγχομαι και σε χώρες οι οποίες είναι and visible ones. Therefore... με απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχει αυτού του είδους ε, η διαφορά. Εμείς προσπαθούμε ε, στις ε, ε, πολιτικές αυτές οι οποίες αφορούν μέτρα τα οποία παίρνουμε μετά από μελέτες επιτόπου να έχουμε μεγάλο βαθμό διαφάνειας και επίσης να παρουσιάσουμε σε όλους την προστιθέμενη αξία που έχει αυτή η δική μας προσέγγιση τέλος ε, η απόφαση, οι αποφάσεις αφορούν εμάς. Ε, ας πούμε ε, το κάναμε και στο Κυργιστάν στην αρχή του χρόνου, το κάνουμε και με την Τινησία, με τον Λίβανο και τις άλλες χώρες οι οποίες προσπαθούν να κινηθούν προς την δημοκρατία αυτό που μάθαμε από όλες αυτές ε, τις ε, καταστάσεις είναι ότι πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στις σωστές δεξιότητες γιατί εμείς δεν θέλουμε να προωθήσουμε στρατηγικές οι οποίες θα μετατρέψουν τους πολίτες σε ρομπότ. Θέλουμε να αναπτυχθεί η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και κατά αυτήν την έννοια ε, βλέπουμε τον σημαντικότατο ρόλο και τη σημαντικότατη θέση που κατέχει η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στη στρατηγική 2020 σε σχέση με το τι κάνουμε και το τι κάναμε στο Κωσυφοπαίδιο και σε άλλες περιοχές του κόσμου ε, και στα πλαίσια της παρουσίας του προγράμματός μας για το 2011 θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως ε, γιατί χρησιμοποιείτε την εργασία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όταν αναφέρεστε στην περιοχή. Είναι γεγονός ότι στο Κωσυφοπαίδιο δίνεται η δυνατότητα συνέχειας δουλεύουμε με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, δουλεύουμε με πολλούς ενδιαφερόμενους ε, και αυτό μας προσδίδει αξιοπιστία. Ιδιαιτέρως δε για το κοσυφοπαίδιο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, ε, να συνεργαζόμαστε με το κεντρικό επίπεδο, με το συμβούλιο αυτό σε κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε όσον αφορά την οικοδόμηση ικανοτήτων, ε, όσον αφορά την σωστή υλοποίηση προγραμμάτων. Το 2011 οι προτεραιότητές μας σε γενικές γραμμές και πέρα και έξω από το κοσυφοπέδιο αφορούν την ανάπτυξη στρατηγικής, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες των αντιστοίχων χωρών. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και χώρες στις οποίες δεν ε, υπάρχουν ιδρύματα ή όργανα που να μετρούν τις ανάγκες της αγοράς. Ε, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χώρες οι οποίες δεν έχουν ακριβώς τα ίδια συστήματα με εμάς. Ε, θα ασχοληθούμε και το 2011 ιδιαιτέρως με την μετανάστευση αλλά ανάποδα, δηλαδή το τι γίνεται όταν επιστρέφουν οι μετανάστες από τις χώρες μετανάστευσης στις ε, πατρίδες τους και αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να, να, αυξηθεί περαιτέρω η μετανάστευση και ο ρυθμός μετανάστευσης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, δημιουργούμε περιφερειακές στρατηγικές όπως ας πούμε αυτή η, περι... στρατηγική για την περιφέρεια του Δουνάβεως και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα, προβλήματα των περιοχών. Ο κύριος Χιμένες, ε, Χουάν Χιμένες ε, Βαλντέ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους και για τις ερωτήσεις, αλλά τον Αλεχάντρο Σέρκας ιδίω να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Σε ευχαριστώ Αλεχάντρο. Σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την κρίση και τον αντίκτυπό τη, έχω να πω ότι ήταν μια από τι προτεραιότητέ μα ε, την τελευταία περίοδο και θα συνεχίσει να είναι, για να δούμε πώ μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τον αντίκτυπο και τι αλλαγέ που έχουν επισυμβεί στη διάρκεια τη κρίση, να προσπαθήσουμε να τι κατανοήσουμε και να δούμε και προ το μέλλον βέβαια, να δούμε μπροστά. Μπορεί να ήρθα από το Δουβλίνο σήμερα, ε, αλλά οι κρίση δεν θα είναι πάντα εδώ και θα πρέπει να δούμε και προς το μέλλον. Και όταν ξεκινήσει η ανάκαμψη θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα και να τα εφαρμόσουμε και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε ό,τι αφορά την ε, απασχόληση των νέων, παραδεχόμαστε και εμείς ότι είναι σαφής προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε και φέτος το έργο που ξεκινήσαμε πέρυσι. Πέρυσι κάναμε μια συγκριτική αναλυτική έκθεση συγκεντρώνοντας πληροφορίες από όλα τα κράτη-μέλη, τις οποίες και συγκρίναμε αναλυτικά και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν εντός του πρώτου τριμήνου. Θέλουμε να συμπληρώσουμε την έκθεση αυτή με ένα νέο σχέδιο που θα επικεντρώνεται στους νέους εκείνους που ούτε είναι στον τομέα της εκπαίδευσης, μάλλον που ούτε είναι σε, κάνουν σπουδές, ούτε έχουν βρει ακόμη θέση εργασίας. Σε ό,τι αφορά την έρευνα, εμείς δεν είμαστε ερευνητικός φορέας ε, αμυγός. Προσπαθούμε να δίνουμε κάποια στοιχεία στους χαράκτες πολιτικής. Και σίγουρα θα κάνουμε και πολλές προσπάθειες στον τομέα της επικοινωνίας. Το 23% του προπολογισμού μας για το 2011 θα, έχει, ε, θα αφιερωθεί ακριβώς στην επικοινωνία. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε μικροί οργανισμοί στο μέγεθος. Δεν έχουμε ανεξάρτητους πόρους. Άρα μας ενδιαφέρουν και κάποιες εκδηλώσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, όπως συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλους φορείς. Για το συγκεκριμένο ζήτημα της ευελιξίας με ασφάλεια, του flexicurity, ναι, πράγματι πρέπει να δούμε τη συνολική δέσμη των διαφορετικών μέτρων που είναι υπό την γενικότερη αυτή ομπρέλα της ευελιξίας με ασφάλεια και να δούμε και το πώ υλοποιείται, πώ εφαρμόζεται στην πράξη η έννοια αυτή και στη διάρκεια τη κρίση. Αυτό που θα κάνουμε φέτο είναι ουσιαστικά να δώσουμε συνέχεια και να συμπληρώσουμε την ανάλυση μετά τις προηγούμενες μας εργασίες και σε επίπεδο του Ιδρύματός μας αλλά και με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναλύσουμε λοιπόν διαφορετικές καλές πρακτικές και πολιτικές θα εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το δημόσιο τομέα και την αποτελεσματικότητά του, είναι ένα γενικότερο θέμα. Δηλαδή, θα αναλύσουμε το θέμα αυτό στο πλαίσιο διαφόρων σχεδίων, αλλά το επίκεντρό μας είναι η κεντρική δημόσια διοίκηση Ίσως θα μπορούσαμε κατά το, στο μέλλον να διευρύνουμε το πεδίο αλλά προς το παρόν θα επικεντρωθούμε εκεί, στο μικρό αυτό κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Ρωμά, είναι ένα ταπεινό, μικρό πρόγραμμα. Μας έδωσε το συγκεκριμένο αυτό αίτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ξεκινήσουμε με μια βιβλιογραφική έρευνα που θα γίνει έτσι στο οργανισμό μας χωρίς να δαπανίσουμε πολλά ποσά και θα επικεντρωθούμε κυρίως στους Ρωμά. Αυτά. Ευχαριστώ. Euh, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριο Κρίστιαν Λετμάιερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Θα ήθελα να απαντήσω το ερώτημα του κυρίου, τα ερωτήματα του κυρίου ε, Σέρκας και της κυρίας Μωράν από κοινού γιατί έχετε δίκιο. Η πρόβλεψη δεξιοτήτων δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν ε, το ε, ανακαλύψαμε ξαφνικά, το εφήβραμε δύο χρόνια πριν. Απλώς αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε έναν μηχανισμό βάσει του οποίου αυτή η πρόβλεψη δεξιοτήτων ε, θα μπορέσει να γίνει ε, ένας, συστηματικ... ένας μηχανισμός συστηματικής μετάδοσης έτσι ώστε να διασυνδεθεί με την αγορά. Ίσως είναι πολλαπλή οι τρόποι ε, με τους ε, οποίους μπορεί κανείς με τρόπο ρεαλιστικό να προχωρήσει στη δημιουργία τέτοιου μηχανισμού και βεβαίως εδώ αναφερόμαστε και στις αρχικές ενδείξεις ε, και δεν αναφερόμαστε μονάχα στους νέους αλλά και στους ενήλικες. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν και τις δημογραφικές προβλέψεις ε, και από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε μία, έναν γυράσκοντα πληθυσμό, μία γυράσκουσα ε, αγορά εργασίας. Προσπαθούμε να περάσουμε, να ξεπεράσουμε μάλλον τα πεπαλαιωμένα συστήματα και επομένως να δούμε προς το μέλλον και η εκπαίδευση ή η κατάρτιση θα είναι κυρίαρχα στοιχεία για το μέλλον. Αλλά όμως δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί για την ώρα όσο μπορούμε. Πρέπει να δούμε και από την πλευρά των αναγκών των ανθρώπων Ποιε είναι οι ανάγκες των ε, ανθρώπων, σε τι αναλογία μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε τις, τα, τα προβλήματα αυτά. και επίσης ε, είναι συντριπτική πλειοψηφία των ε, ατόμων με χαμηλά προσόντα. Ε, βεβαίως μειώθηκε λίγο ο αριθμός τους, αλλά παρόλα αυτά είναι η συντριπτική πλειοψηφία και επομένως προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε, προς τα εκεί το Σεντεφόπ στρέφεται έτσι ώστε να προσπαθήσει να δει ε, τι πρέπει να γίνει, τι έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στον τομέα αυτό ήδη και τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε στο μέλλον τα πράγματα να είναι καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Μπάουρ και για την δικιά σας ε, ερώτηση. Πρέπει να ζητήσω και κατά κάποιο τρόπο συγγνώμη γιατί ε, αυτό που αναφέρεται είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή τα, συγκεκριμένα προσόντα, τα, οι συγκεκριμένες δεξιότητες ε, μπορεί να αφορούν μονάχα μια συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως θα πρέπει ε, να έχουμε τη δυνατότητα να ε, βρούμε τις δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τις περιφέρειες, με τις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες. Αυτό δυστυχώς το ΣΕΝΤΕΦΟΠ δεν μπορεί να το, να το κάνει. Δεν είναι δυνατόν το ΣΕΝΤΕΦΟΠ να κατέβει σε τέτοιο βαθμό ε, λεπτομέρειας. Επίσης, ε, όσον αφορά τη, την επόμενη ερώτησή σας, είναι γεγονός ότι συμμετέχει το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, αλλά είναι καταρχήν μια εργασία της Γενικής Διεύθυνσης ε, Απασχόλησης και βεβαίως όλες αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες στρατηγίες, συγκεκριμένα μέτρα από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών, αυτές οι οποίες θα παρέμουν σε περιφερειακό επίπεδο και εάν τα συστήματα αυτά ε, λειτουργήσουν καλά τότε κυρίω θα είναι θέματα τη κεντρικής κυβέρνηση και επιτυχία των κεντρικών κυβερνήσεων και όχι του ΣΕΝΤΕΦΟΠ παρότι θα θέλαμε να είμαστε και πιο παρόντε. Ο κύριος Τάκαλα, τελευταίος ε, ομιλητής. <clears throat> Um, I start from the... Uh, σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από τα σχόλια του Αλεσάνδρου και της ε, κυρίας Σαλτιέ. Σας ευχαριστώ καταρχήν όλους για τα ενθαρρυντικά σας λόγια και χαίρομαι που είστε ικανοποιημένοι από το έργο που σας παρουσιάζουμε. Ε, γιατί ε, έχουμε καταστάσεις ε, αναπηρίας σε άτομα πολύ νεαρά, ακόμη και 32 ετών. Είναι ένα φαινόμενο που πολύ συχνά το παρατηρούμε. Μπορεί μία εργαζόμενη να έχει πολύ καλές επιδόσεις και στο σχολείο και, στις, και στην επαγγελματική της σταδιοδρομία. Ακούει αυτά τα οποία της λέει ο εργοδότης και συνεχώς κάνει όλο και περισσότερα, προσφέρει όλο και περισσότερα μέχρι που εξαντλείται και φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να παράγει, εξαντλείται και αναγκάζεται να αποχωρήσει από το χώρο εργασίας. Και αν δούμε τις ε, αναπηρίες και τους βασικούς λόγους, ε, οι βασικοί λόγοι είναι η μείωση σκελετικές διαταραχές και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που είναι και οι πιο δαπανηροί. Τα τρία τέταρτα των δαπανών για πρόορη συνταξιοδότητη οφείλονται σε τέτοια προβλήματα. Για να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτό θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την ηλικία των 65 ή των 67 ή των 68 όσο θα πούμε, δεν πρέπει να αρχίσουμε τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων όταν θα έχουν ήδη φτάσει στην ηλικία των 50 ετών γιατί τότε θα έχουν ήδη τα μυοσκελετικά προβλήματα ή τις ψυχικές διαταραχές και δεν θα θέλουν να εργαστούν άλλο. Θα πρέπει πολύ νωρίτερα να αρχίσει η διαχείριση αυτών των προβλημάτων αυτό που ρώτησε η κυρία Μπάουε για τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για αυτά τα θέματα που ανέφερα, τις μειοσκελετικές διαταραχές ε, και τους ε, ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, οι γυναίκες φύγονται ε, περισσότερο από τους άνδρες και στα δύο αυτά προβλήματα είναι περισσότερο ευάλωτες οι γυναίκες. Όχι γιατί είναι πιο αδύναμες οι γυναίκες, αλλά διότι συνήθως οι γυναίκες θέλουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, θέλουν να προσφέρουν περισσότερα και γι' αυτό ε, καταλήγουν σε αρνητικές συνέπειες. Ε, για το θέμα των νομικών απαιτήσεων και για τα προληπτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε. Το πρώτο είναι, το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τους υφιστάμενους κανονισμούς Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών τα οποία ισχύουν βάσει των κανονισμών και αυτών τα οποία εφαρμόζονται στην πράξη. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε στη διάθεσή μας και να ακολουθήσουμε και τη Σύμβαση 187 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Χρειαζόμαστε τα νομικά μέσα που θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας, μοντέλα κατάρτισης, καλές πρακτικές καθώς και μέτρα επιβολής της νομοθεσίας. Δεν είναι εύκολο να έχουμε νομικά μέσα για να ε, εμποδίσουμε τα προβλήματα που οφείλονται στο στρες. Μπορούμε όμως ε, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προληπτικά για θέματα όπως είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές, ε, ο καρκίνος, άκουσα ένα ερώτημα σχετικά με αυτό, είναι θέματα ε, στα οποία μπορούν οι νομικές διατάξεις να βοηθήσουν στην πρόληψη. Αυτό το οποίο δεν είναι σωστά οργανωμένο από νομική πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών. Γιατί θα έπρεπε να έχουμε επιτόπου νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολογική υποστήριξη, που άνθρωποι που είναι ειδικοί στον ε, τομέα των ε, ε, ιατρικών υπηρεσιών που θα συνεργάζονται υπέρ της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών. Σε ορισμένε πρώην σοσιαλιστικέ χώρε υπήρχαν κάποια συστήματα τα οποία διαλύθηκαν και έχουμε φτάσει να μην υπάρχει καθόλου προστασία σήμερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα των όσων θα μπορούσαν να γίνουν για την πρόληψη. Και θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε αυτά τα μέτρα στον χώρο εργασίας. Για την ερώτηση που ε, υπέβαλε ο Ιρλανδός Ευρωβουλευτής ε, σχετικά με την τάση να υπάρχουν όλο και περισσότερα ατυχήματα στη γεωργία. Νομίζω ότι τα ατυχήματα στον τομέα της γεωργίας οφείλονται στη βιομηχανοποίηση της ε, γεωργίας. Όλο και λιγότερα άτομα κάνουν περισσότερες εργασίες, περισσότερα μεγαλύτερη ισχύ των γεωργικών ελκυστήρων, περισσότερα μηχανήματα και καμιά φορά χωρίς καμία καθοδήγηση αφήνουμε τους ε, εργαζόμενους ε, να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενοι που δεν έχουν καμία πληροφόρηση, καμία ενημέρωση, δεν γνωρίζουν καθόλου τα μέτρα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν και γι' αυτό εκτίθεται σε μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Α, και κάτι ακόμη. Είναι η τελευταία φορά που εμφανίζομαι εδώ γιατί σε ένα χρόνο από τώρα θα έχω συνταξιδοτηθεί ήδη. Σας ευχαριστούμε και τους τέσσερις καλωσορίζουμε κάποιους, αποχαιρετούμε κάποιους άλλους. Ε, για μας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επαφές που έχουμε μαζί σας. Είναι ποικίλα τα θέματα και παίρνουμε μεγάλο πλούτο εμπειριών. Όλα τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε για μας είναι πολύτιμα. Ακούσαμε αυτό που είπε ο σας Δερόσα για τα ατυχήματα στον γεωργικό τομέα και θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε με τα θέματα στρες και με τα στατιστικά στοιχεία από τη Γαλλία όπου στο γεωργικό τομέα υπάρχουν πολλές ανησυχίες, περισσότερες ανησυχίες από ό,τι τα περασμένα χρόνια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση όμως. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στη χρονιά να επισκεφθούμε και το Μπιλμπάο και το Δουβλίνο. Και από την εμπειρία μου στο Τωρίνο Μπορώ να πω ότι είναι πολύτιμες αυτές οι επισκέψεις επιτόπου. Θα σας επισκεφθούμε λοιπόν και νομίζω ότι και για σας είναι σημαντικές αυτές οι επισκέψεις γιατί μπορείτε να μας δείξετε πολύ περισσότερο εμπεριστατωμένα τη δουλειά που κάνετε. Όλα στην προοπτική του Ευρωπαϊκού Ιδεόδους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία που είχαμε για την ανταλλαγή εμπειριών. Σας εύχομαι καλή δουλειά μέσα στο 2011 γιατί είναι πολλά τα θέματα στα οποία είστε οι εμπειρογνώμονές μας και όπου χρειαζόμαστε την εμπειρία σας για να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο και το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Σας ευχαριστούμε. Euh, Θα δώσω τώρα τον ε, λόγο στον κύριο Ορί για την ε, παρουσίαση της πρώτης απαλλαγής Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα 3 και θα πρέπει να του ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω για λίγο. Θα πάω σε μια άλλη επιτροπή και θα δώσω τον λόγο στην την Προεδρία στην Αντιπρόεδρο. Κύριε Ορή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο. Okay. uh... Ωραία, να ξαναρχίσω λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδίνετε το λόγο ως νέα προεδρεύουσα. Την τελευταία φορά είχαμε ήδη αναφερθεί ε, στις απαλλαγές ε, διαφόρων ε, κέντρων και ιδρυμάτων και είχαμε τότε διαπιστώσει ότι όλο και λιγότερα προβλήματα έχουμε. Υπάρχουν όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα επί των οποίων όμως έχουμε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορούμε να τα εξουδετερώσουμε τα προβλήματα αυτά, να τα επιλύσουμε. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε πολλά σε αυτά που έχουν ήδη προταθεί. Κάποιες ε, τροπολογίες μονάχα έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι και ε, θα ασχοληθώ με όλες τις ε, με όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς από κοινού. Όσον αφορά τις τροπολογίες, ναι, ναι, ναι, είχαμε πει ναι, το, ε, είχαμε προβλέψει ότι θα μιλήσετε για όλες τις απαλλαγές και μετά θα μιλήσουν και οι σκιώδεις ηγητές ε, πάλι για όλα. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Επομένως υπάρχουν ε, κάποιες τροπολογίες τις οποίες θα ήθελα να αναφέρω. Ε, κάποιες γλωσσικές ε, κυρίως διορθώσεις. Μπορώ να δεχτώ τις τροπολογίες αυτές. Μπορώ να δεχτώ λοιπόν όλες τις τροπολογίες εκτός από την τροπολογία Obermeier που απαιτεί γιατί κάποιες ε, προσωπικές αναφορές για, ε, για το Δουβλίνο, για το Ίδρυμα του Δουβλίνου. Νομίζω ότι ήδη βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Τα προβλήματα αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν ξεπεραστεί ε, και νομίζω ότι και σε προσωπικό επίπεδο και οι επιπτώσεις ήταν σαφείς. Ε, ήδη, ήδη έχει ξεκινήσει να διαφύνεται η λύση και επομένως θεωρώ ανώφελο να στηρίξουμε την τροπολογία αυτή. Πέραν αυτών όλες οι αποσαφηνήσεις ε, που δίνονται από τους σοσιαλιστές ε, είναι αποδεκτές και τις δέχομαι και εγώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Επομένως σε λίγο μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Ρέο, κύριο Τσάκας. Μετά κυρία Πέρες. Ο κύριος Σέρκα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συνάδελφός μου, Κίνγκα Γκέντς, υποτίθεται ότι θα ήταν εδώ, γιατί με τον κύριο Τσάμπα Όρη ο Σκιώδης εισηγήτρια παρακολούθησε την εκπόνηση των εκθέσεων αυτών αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι και δύσκολο να την υποκαταστήσω, διότι η Σοσιαλιστική Ομάδα συμφωνεί πλήρως με το έργο που έχει επιτελέσει ο κύριος Όρη. Συμφωνούμε με τις τροπολογίες που δέχεται, αλλά και με αυτές που δεν δέχεται. Και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ήταν ιδιαίτερα γενερόδωρος, δέχτηκε τις τροπολογίες της Σοσιαλιστικής Ομάδας, άρα η δική μου ομάδα συμφωνεί απόλυτα με το έργο του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σέρκας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρου τη Μάριαν Χάρκιν, τη συναδέλφου, θέλω να λάβω το λόγο. Εκείνη είναι η σκιώδη εισηγήτρια. Συμφωνεί με το σχέδιο γνωμοδότηση που τονίζει τα βασικά θέματα, όπω είναι η ανάγκη βελτίωση τη ε, οικονομική διαχείριση και τη μείωση του εσωτερικού του κόστου εργασία. Ε, την προσπάθεια της Επιτροπής ε, να ληφθούν υπόψη ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και οι συνοπτικές ετήσιες εκθέσεις. Το σχέδιο γνωμοδότησης τονίζει την ε, τρέχουσα κατάσταση και τις ανησυχίες που υπάρχουν ε, στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και μιλάει για τα ε, βήματα πρέπει να ληφθούν για να συμμορφωθούμε με τα ζητήματα που δείτε από το ελεγκτικό συνέδριο. Ακόμη η σχεδόν δεν υποστηρίζει την πρώτη τροπολογία. Υπάρχουν λόγια για τη μεταφορά. Η δεύτερη τροπολογία είναι γλωσσική φύσεω. Για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρόμοια σχόλια όπω και για το Ίδρυμα για ε, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία χαιρετίζει τη δέσμευση του Ιδρύματος ε, να ερμηνεύσει αυστηρά ε, τον, οικονομικό, δημοσιονομικό κανονισμό και τη δέσμευσή του να ε, γίνουν πιο αυστηρές οι μεταφορές ποσών. Πρέπει να εξηγηθούν καλύτερα οι λειτουργίες του οργανισμού ε, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ τώρα και πάλι το σχέδιο γνωμοδότησης ε, έχει καταρτιστεί ε, σωστά. Τονίζει τα θέματα τα οποία τονίζουν και από το ελεγκτικό συνέδριο. Η δεύτερη τροπολογία δεν είναι κέρια σημασία, βελτιστοποίηση αντί μεγιστοποίηση. Επίσης πιστεύει ότι μας δίδονται πληροφορίες για το μελλοντικό ρόλο του οργανισμού. Για το ε, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης στην πρώτη τροπολογία πιστεύει η Σκιώδης Συγγήτρια ότι αυτό που λέμε για τη λογοδοσία είναι πολύ ευρύ ποιες είναι οι συνέπειες αυτού που λέμε. Όταν μιλάμε για το προσωπικό, μιλάμε για όλα τα επίπεδα του προσωπικού. Αυτό είναι ένα ερώτημα της κοιόδους συγγήτριας. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες ε, για το προσωπικό. Πάντως, γενικά δεν υποστηρίζει την τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο. Θα δώσω και πάλι λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Όρη. Επομένως, Νομίζω ότι ήταν σαφές το περιεχόμενο των τροπολογιών, έτσι ακριβώς όπως το σχολίασαν και οι συνάδελφοι που μόλις πήραν το λόγο. Ε, ακούσαμε την ε, τροπολογία που αφορά την, ε, μία, το, ένα ίδρυμα, έστω και αν αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, μπορούμε να το ψηφίσουμε. Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων εδώ και των οργανισμών οπωσδήποτε έχουν ε, ε, πάρει όλα τα θετικά στοιχεία της ε, εργασίας που έχουμε κάνει και της ε, συζήτησης που κάναμε εδώ. Δηλαδή ε, το νόημα είναι ότι εμείς ε, διαφορόμαστε πάρα πολύ για την εργασία τους, την αξιολογούμε πολύ θετικά και θέλουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης εισηγητάς, κυρίως δε την Έρικα Σούλτς για την βοήθειά τους και νομίζω ότι τώρα πια είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε το, τη γνωμοδότηση αύριο. Ευχαριστούμε κύριε Ορή. 1η Φεβρουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2010. Η συγκίτρια η κυρία Νάντια Χίρς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάναμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή τη γνωμοδότηση και υπάρχουν πολλές τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και όλους εκείνους που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε ορισμένα θέματα και να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Κάποιες τροπολογίες τις ομαδοποιήσαμε και έχω και τη συμφωνία ε, κάποιων συναδέλφων. Ε, ελπίζω ότι οι περισσότερες συμβιβαστικές τροπολογίες, πολλές τουλάχιστον από αυτές τις τροπολογίες, θα έχουν συνοψίσει σωστά τις ανησυχίες μας για τα θέματα της φροντίδας των παιδιών, για τα θέματα της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων, τι μπορεί να γίνει δηλαδή για να έχουμε συμφιλίωση της εργασίας με την προσωπική ζωή. Νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε σωστές συμβιβαστικέ λύσεις. Ένα σημαντικό σημείο ε, αφορά και τα υποχρεωτικά, τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις για διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να έχουμε εθελοντικές ε, ποσοστώσεις ή υποχρεωτικές ποσοστώσεις. Είναι θέματα ε, ε, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα. Υπάρχει το θέμα το οποίο συζητείται και στην ε, ε, Κοινωνική Επιτροπή, το θέμα της ε, απασχόλησης για όλους, ιδίως η απασχόληση για τις γυναίκες και τις νέες κοπέλες και ιδίως μετανάστριες. και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Επιτροπή Γυναικών και θα φανεί και στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Άντια Χίρς. Jutta Steinrück, Thomas Mann, Λόπε Φοντάνια, Jutta Steinrück καταρχήν. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Χίχς και να την ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μερικές φορές και την τελευταία στιγμή καταφέραμε να συνεννοηθούμε για ε, κάποια θέματα. Θέματα που ήταν για μας ε, σημαντικά ήταν ότι θέλουμε να προωθήσουμε την ε, ισότητα και να κάνουμε ορισμένα θέματα υποχρεωτικά και δεσμευτικά. Γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές διακήρυξη προθέσεων μέσα στα περασμένα χρόνια χωρίς αποτελέσματα και με την κρίση φάνηκε ότι οι γυναίκες εθίγησαν περισσότερο. Γι' αυτό καλό θα ήταν να μπουν κάποιες δεσμευτικές διατάξεις στον α ή στο β τομέα, όπως παραδείγματος χάρη για ποσοστώσεις, για διευθυντικές θέσεις, για θέσεις τελεχών για γυναίκες ή για διοικητικά συμβούλια. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία ε, από τη Βελική Προεδρία και μιλάμε για ε, δείκτες απασχόλησης για τις ε, γυναίκες όπου θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Είναι ένα θέμα που και ο Υπουργός είχε τονίσει στην Επιτροπή μας. Πρέπει να βελτιώσουμε τη θέση των γυναικών, ιδίω σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Εδώ υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και το θέμα του gender budgeting, κατάρτιση του προπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου δηλαδή, είναι ένα θέμα που πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη. Έχω και μία ερώτηση για τις τροπολογίες 42 και 43. Ίσως να είναι γλωσσικό το πρόβλημα και να οφείλεται στη μετάφραση. Θα μπορούσαν οι συντάκτες της τροπολογίας να μας εξηγήσουν περί την Για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Τόμας Μαν και μετά η κυρία Λόπε Φαντάνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την Άντια Χίρς. Έχουμε τρεις προτάσεις συμβιβαστικών λύσεων, α, β και γ και ζήτησα από την πολιτική μας ομάδα και τις τρεις συμβαστικές λύσεις να τις υποστηρίξει γιατί νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ καλή λύση. Διαφωνείτε με την ε, τροπολογία 9 ε, σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ε, άδεια του, της μητέρας και του πατέρα. Στο θέμα της προστασίας της μητέρας πάντοτε έχουμε συζητήσει τα θέματα διαφορών που υπάρχουν και νομίζω ότι χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση τέτοιων διατάξεων για να έχουμε κάτι πιο προσεκτικό και να έχουμε αποτελέσματα με τα οποία θα μπορούσαμε να είμαστε σύμφωνοι. Και για την 26, την οποία επίσης ε, απορρίπτει η συγγήτρια ε, για τις νομοθετικές ε, προτάσεις, πιστεύω ότι εδώ έχουμε ένα σημαντικό θέμα και δεν συμφωνώ με την συνάδελφο Κορνέλισεν. Ε, για την 35 υπάρχει κάποια αντίφαση, γιατί νομίζω ότι εδώ οι σοσιαλιστές λένε ότι θέλουμε ε, να έχουμε σχέδια τα οποία θα είναι νομικά εδρεωμένα, αλλά όταν κάτι ε, ξεκινάει από τους κοινωνικούς εταίρους δεν είναι σαφές πώς θα προκύψει αυτό γιατί αν θέλουμε να έχουμε ανεξαρτησία των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να είναι στα χέρια τους. Γι' αυτό υπάρχουν εξάλλου κοινωνικοί εταίροι και έχουν επαρκή εμπειρία και δεν αρκεί να πούμε ότι σε ορισμένα θέματα θα έχουμε ε, δυνατότητα παρέμβαση και σε άλλα όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να, με αυτά τα μέσα να νομιμοποιούμε και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων για την 53 υπήρχαν προβλήματα με τις μεταφράσεις σε κάποιες γλώσσες. Λέμε απορρίπτει τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις για τα διοικητικά και τα υποπτικά συμβούλια. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική υποστήριξη για αυτό το θέμα για μένα είναι ένας τομέας ιδιαίτερα σημαντικός. Και στην τροπολογία 58 της κυρίας Φιγκερέιντο για τις διακριτικές μεταχειρήσεις ε, όσον αφορά τις, μισθολο... τις μισθολογικές διακρίσεις. Ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρη θέση η οποία λήφθη σε σχέση με την ε, γνωμοδότηση αυτή με την ε, τροπολογία συγγνώμη αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Τομασμάν, η κυρία Λόπες Φοντάνια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Νομίζω ότι ο σύντροφό μου Τόμα Μαν έθιξε όλα τα θέματα. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Χίρς. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο να εργάζεται κανείς μαζί της Ξέρετε, όλοι περίπου τις ίδιες θέσεις έχουμε και τον ίδιο στόχο, δηλαδή επιτέλους να πετύχουμε σιγά σιγά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και νομίζω ότι πρακτικά έχουμε καταλήξει σε συμφωνία ε, επί του συνόλου των ε, τροπολογιών με εξαίρεση τα άρθρα για τις ποσοστώσεις που και στη δική μου πολιτική ομάδα δεν έχουμε ακόμη συνένεση και στο Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξανασυζητήσουμε αν γίνεται. πάντω, ούτω ή άλλω θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Στρέλα και η κυρία Μπάουερ έχουν ζητήσει το λόγο. κυρία Μπάουερ και μετά η Γιούτα Στάινουρικ άλλη μια φορά. Η κυρία Στρέλα πρώτα, συγγνώμη, η κυρία Στρέλα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτά που ανέφερε συνάδελφος Στάινρουκ και να πω ότι συμφωνούμε όλοι επί των στόχων αλλά όχι αναγκαστικά επί των μέσων που θα χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους. και ορισμένες τροπολογίες προτείνουν διαφορετικά μέσα. Ιδίως για το στόχο της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη συνεισφορά στην ανάπτυξη, όπως ορίζεται στη στρατηγική για το 2020. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους την πρωτοβουλία της συντηρητικής νορβηγικής κυβέρνησης που όρισε ποσοστώσεις για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η βασική ιδέα δεν ήταν η πρόθεση της ισότητας των φύλων, κυρίως οικονομική ήταν η λόγη. διότι υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που δείχνουν ότι η συμμετοχή γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο οδήγησε τις εταιρείες σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Η εταιρεία Catalyst έχει κάνει μια μελέτη που δείχνει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων εταιριών οδήγησε σε αύξηση κατά 73% της χρηματιστηριακής αξίας των εταιριών. Η ιδέα λοιπόν του να μπει μια τέτοια ποσόστοση έχει σαφώς θετικές επιπτώσεις και αυξάνει τη συμμετοχή των γυναικών αλλά έχει και θετικές οικονομικές επιπτώσεις. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι διότι στη γνωμοδότηση δίνεται ιδέουσα βαρύτητα στη δημιουργία δομών φροντίδας των παιδιών, παιδικών σταθμών παραδείγματος χάριν, όπως επίσης και στην ιδέα της συμφιλίωσης της επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Ο κύριος λόγος που φεύγουν από την αγορά εργασίας οι γυναίκες είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα του ότι δεν μπορούν να συμφιλιώσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τη δική μου έκθεση σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Στην οδηγία αυτή συμπεριλαμβάνονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Δεν έχουμε βέβαια ακόμη την συμφωνία του Συμβουλίου. Αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν τη θέση του Κοινοβουλίου. Έχουμε την δική μας θέση για την γονεϊκή άδεια και αναθεωρείται η σχετική οδηγία. Και έχουν συμπεριληφθεί και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων. η νομοθεσία που ήδη ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αυτά τα οποία ήδη έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να αγνοηθούν από το Συμβούλιο. Ακόμη θέλω να αναφέρω κάτι για την τροπολογία 28 για την διαφορά αμοιβών που δεν είναι πια 15% αλλά 18%. Άρα εδώ δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν επιδεινωθεί και ανέρχονται σε 28%. Πρέπει να το διορθώσουμε λοιπόν το ποσοστό που αναγράφεται εκεί. Επίσης στην τροπολογία 4 όπου αναφέρονται οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας πρέπει να πούμε ότι η στρατηγική αυτή έληξε το 2010 και πρέπει πλέον να μιλάμε για τους στόχους της στρατηγικής για το 2020. Σε αυτό πρέπει να αποσκοπούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Στρέλα. Η κυρία Μπάουερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι λίγο περίεργο που η κυρία Εστρέλε είπε τα μισά τουλάχιστον από αυτά που ήθελα να σας πω. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να θίξουμε το ακόλουθο ζήτημα. Η στρατηγική 2020 και οι στόχοι που αφορούν την απασχόληση δεν θα υλοποιηθούν παρά με την προϋπόθεση να δημιουργηθεί μία, ε, ένα υπόβαθρο όσον αφορά τις υπηρεσίες. Γιατί όσον αφορά τις γυναίκες ξέρουμε ότι έχουμε μία αύξηση κατά 20% της απασχόλησης, εάν δεν δημιουργηθούν υπηρεσίες, όπως ας πούμε ε, παροχή ε, παροχή, ε, βοήθεια όσον αφορά τα παιδιά, ε, ε, σημεία φύλαξη των παιδιών, υποδομές για, για τους ηλικιωμένους, τότε δεν θα μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να δουλέψουν. Με αυτή την έννοια έχουμε υποβάλει και την τροπολογία 28 και επίσης η Επιτροπή πρέπει να μας δώσει σαφή απάντηση όσον αφορά την ε, ε, διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Γιατί αυτή η διάσταση, αυτή η διαφορά διαρκώς μεγαλώνει. Για κάποια μικρή περίοδο ε, έκλεινε κάπως η ψαλίδα, αλλά τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε ότι ξανανοίγει η ψαλίδα και μεγαλώνει η διαφορά. Η Κομισιόν δεν μας έχει απαντήσει ακόμα το Κοινοβούλιο έκανε κάποιες νομοθετικές προτάσεις, ούτε για αυτές έχει κάποια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν βλέπουμε να αναλαμβάνει και πολύ ενεργητικό ρόλο. Εμείς κάνουμε συστάσεις. Αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Κάθε χρόνο κάνουμε εκθέσεις για την θέση των γυναικών. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έστω και εάν πρέπει να ε, επανενεργοποιήσουμε κάποιες παλιές προτάσεις ε, παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε και καινούριες ε, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και όχι πάντα προς το καλύτερο. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Στάινρουκ για να απαντήσει. Εν συντομία, μετά τις παρατηρήσεις του Τόμας Μαν σχετικά με την τροπολογία 35. Έχουμε, εμείς ε, προσανατολιστήκαμε στο ισπανικό παράδειγμα μέσω μιας δεσμευτικής νομοθεσίας και μέσω της εφαρμογής από τους κοινωνικούς εταίρους βελτιώθηκε η συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Αυτή ήταν η κατεύθυνσή μας και γι' αυτό αναφέραμε τα παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ευρώπη. Αλλά μπορούμε να το εξηγήσουμε λεπτομερέστερα αν θέλετε. Νομίζω ότι ήταν καλό παράδειγμα και χρήσιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητάει το λόγο. Η Νάντια Χίξ, ε, που είναι η συγγήτρια, έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Το θέμα των σχεδίων πρόθεσης της ισότητας θα έχουμε συζητήσει διμερώς και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Τόμας Μαν που και αυτός μίλησε για το θέμα αυτό δεν είναι ξεκάθαρο πώς μπορούμε να εδραιώσουμε αυτές τις πρακτικές σε νομοθετικά μέσα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι το γραφειοκρατικό και γι' αυτό με προσοχή το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Έχετε δίκιο, πρέπει να διορθώσουμε το ποσοστό. Δεν είναι 15 αλλά 18% δυστυχώς. Είναι μεγαλύτερη διαφορά μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών για την τροπολογία 4 το θέμα ε, των εθελοντικών ποσοστώσεων είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε ακόμη. Νομίζω από αυτά που έχουμε συζητήσει η εντύπωση που προέκυψε ότι υπήρχαν σαφώς ξεκάθαρες θέσεις. Ξέραμε τα επιχειρήματα τα οποία αντιλάγησαν και νομίζω ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαφέρουν κατά πολύ τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών και είναι διαφορετικές οι αξιολογήσεις κράτος μέλος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να καταλήξουμε σε καλύτερη συμβαστική λύση από αυτού. Για την τροπολογία 34 της Γιούτα Στάνρουκ, ε, συμφωνήσαμε για μια προφορική τροπολογία, για να συμπληρώσουμε αυτή την τροπολογία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν ε, το αν είναι δίκαια τα φορολογικά τους ε, συστήματα και αν δίδονται επαρκή φορολογικά κίνητρα. Η τωρινή διατύπωση θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι έχει φορολογικές αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό με την προφορική τροπολογία που ε, συμφωνήσαμε να κάνουμε, θα λέμε ότι ε, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τα φορολογικά του συστήματα για να δουν αν μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Και με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα μπορούν να συμφωνήσουν. Ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ αυτής της έκθεσης για να μπορέσουμε να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Άντια Χίρς. Η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο. Γιατί μεθαύριο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Γυναικών. Αυτά λοιπόν για το σημείο αυτό. Yeah. Nein, jetzt. Η Νάντια Χίρς είναι η συγγήτρια και για το επόμενο σημείο, το σημείο 12, Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Υποστήριξη Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Νάντια Χίρς, και πάλι λοιπόν. Υπήρχε στην ημερήσια διάταξη το εμβόλυμο σημείο για την ενσωμάτωση των Ρωμά, αλλά τροποποιήθηκε η ημερήσια διάταξη, οπότε έχω εγώ δύο σημεία το ένα μετά το άλλο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ και τον πιο Εισηγητή για τη συνεργασία που είχαμε. Έχουμε κάνει αρκετέ συναντήσει επί του θέματο. Ε, γιατί θέλαμε να καταλήξουμε σε κοινή άποψη και νομίζω τελικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες κυρίως για την ανεργία των νέων υπάρχουν πολλές τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική τροπολογία. Γιατί ακριβώς σε αυτό τον τομέα υπάρχουν πολλές τροπολογίες και πρέπει να βελτιώσουμε κάπως τη διατύπωση. Επειδή είναι και πολύ επίγον αυτό το θέμα, είναι ιδιαίτερα πιεστικό το θέμα της ανεργίας των νέων, πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική τροπολογία. και στην έκθεση αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Πρέπει δηλαδή οι νέοι να είναι σωστά προετοιμασμένοι για την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Ένα θέμα που έχει, είναι, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ανεργία των νέων. Και εδώ είχαμε αρκετέ τροπολογίες αλλά νομίζω ότι θα βρούμε τη σωστή συμβαστική λύση για τις τροπολογίες αυτές. Για το θέμα της χρηματοδότησης επίσης υπάρχουν κάποια σχόλια. Ιδιαίτερα αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προετοιμασία των νέων ε, και των ε, μεταναστών για να μπορέσουν με στοχευμένο τρόπο να χρησιμοποιήσουν το Κοινωνικό Ταμείο για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία, συνεργασία μεταξύ σχολείων, μεταξύ επιχειρήσεων ε, και με την υπηρεσία που ε, παρέχει στους νέους αυτά τα οποία χρειάζονται, όλοι αυτοί θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να μπορέσουν ως τελικό αποτέλεσμα ε, να βοηθήσουν τους νέους να έχουν θέση απασχόλησης για την επαγγελματική κατάρτιση τονίζουμε τη σημασία της ποιότητας και νομίζω ότι και πολλές τροπολογίες ε, αποσκοπούν σε αυτό. Τονίζουμε ε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ε, και το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας. Αυτές είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να τις αναφέρουμε, να τις τονίσουμε και να δείξουμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο και θέλουμε να συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι το βασικό σημείο. Σχέση μεταξύ επαγγελματικής ε, ε, κατάρτισης και πανεπιστημίων είναι άλλο ένα σημαντικό θέμα. Η επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι ένα αδιέξοδο αυτός ο οποίος έχει περάσει από ένα στάδιο επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ε, να περάσει σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Γι' αυτό χρειάζεται ε, ένα, μια σαφή σύνδεση μεταξύ των δύο τομέων. Είχαμε αρκετέ τροπολογίε και για το θέμα τη σύνδεση λοιπόν επαγγελματική κατάρτιση ε, και ανώτατη εκπαίδευση. Θα προσπαθήσουμε να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και η σχέση με την ανεργία των νέων, όπου ίσως χρειάζεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να τονίσουμε τη σημασία του θέματος. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία που έχω σημειώσει. Θα συζητήσουμε με τους κοιόδης της της τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει όλων ούτως ώστε με την έκθεση αυτή να τονίσουμε τα ενδιαφέροντα και των μικρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση. Ευχαριστώ την Άντια Χίρς. Δύο μιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Τσιλέσκα Κύριε Τσιλέσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα να πάρω το λόγο εξ ονόματος του κυρίου Κοσλόφσκι, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής από το ΕΛΚΑ και δυστυχώς δεν είναι εδώ. Έμεινε στην Πολωνία και δεν μπόρεσε να έρθει λόγω ε, σοβαρών χιονοπτώσεων στην Πολωνία. Είναι λοιπόν σκιώδης εισηγητής ε, στην έκθεση της κυρίας Χίρς ε, και ως σκιώδης εισηγητής θα ήθελα να ευχαριστήσει την κυρία Χίρς για την επικοδομητική συνεργασία επί της εκθέσεως για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την υποστήριξη της Δυτικής Ευρώπη 2020. Λαμβάνει υπόψη η έκθεση όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την επαγγελματική κατάρτιση ε, και εκπαίδευση και που είναι βεβαίως απαραίτητα έτσι ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Ο κ. Κοσλόφσκι είναι πολύ ευτυχής με την εξέλιξη της ε, συζήτησης αυτής και έχει υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες τις οποίες θα παρουσιάσω σύντομα εν συντομία μάλλον ε, οι τροπολογίες του απλώς ήθελαν να αποσαφηνίσουν κάποια στοιχεία της εκθέσεως Χίρς ή σε ορισμένες περιπτώσεις να παρουσιάσουν μια άλλη οπτική κάποιων στοιχείων χωρίς να αλλάξει όμως ε, η γενική οπτική. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να είναι απαραίτητα στοιχεία της ε, αγοράς που αλλάζει διαρκώς από κοινωνική και οικονομική άποψη. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να γίνει πιο ευέλικτο. Τροπολογία υπαριθμών 30. Εδώ υπάρχει ένα λάθος μεταφραστικό στην πολωνική εκδοχή. Αντί για διαχείριση έχει ε, εσφαλμένα επιλεγεί η λέξη κατεύθυνση. Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αξιολόγηση των ε, καταρτήσεων έτσι ώστε η κατάρτιση και τα προγράμματα κατάρτισης να είναι υψηλού επίπεδου και υψηλής ε, ποιότητος έτσι ώστε ε, και αυτό αναφέρεται στην τροπολογία 112. Ο κύριος Κοσλόφσκι πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ε, μάθει η κοινή γνώμη ε, να αντιμετωπίζει καλύτερα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ε, η κοινή γνώμη λοιπόν να κατανοήσει ότι η διαβίου εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Τροπολογίες 38 και 45 έτσι ώστε να διασφαλιστεί υψηλής ποιότητας κατάρτιση από την αρχή του κύκλου της κατάρτισης. Για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί και η έννοια των ε, κυρίων προσόντων, κάποιων προσόντων ε, που θα παίζουν ρόλο κλειδί σε ολόκληρο το σύστημα κατάρτισης και το αναφέρουμε αυτό στην ε, συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι όσον αφορά την επαγγελματική ε, κατάρτιση πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, σε συστήματα κινήτρων και όχι σε υπερβολικά αυστηρό έλεγχο. Ο κύριος Κοσλόφσκι λοιπόν προτείνει επαναδιατύπωση της παραγράφου 5 όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί στην πρόταση, στην παράγραφο έτσι όπως την προτείνει η κυρία Χίρς, ε, δίνεται η αίσθηση ότι μέσω ελέγχου ποσοστώσεων, συμμετοχής γυναικών κτλ. Ε, γίνεται μια προσπάθεια υπερβολικού ελέγχου του αριθμού ανδρών και γυναικών. Ο κύριος Κουσλόφσκι επίσης θα ήθελε να εντάξει στην έκθεση Ε, κάποιες ε, εκκλήσεις ε, προς τα κράτη-μέλη έτσι ώστε αυτά να λάβουν υπόψη τους την ισότητα των ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Τροπολογία 70 εκεί υπογραμμίζεται η σημασία των ε, κοινωνικών εταιρικών σχέσεων, ε, τις σχέσεις ε, με την τοπική διακυβέρνηση, συνδικάτα κτλ. έτσι ώστε η επαγγελματική κατάρτιση να διασυνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς. Οι άλλες τροπολογίες του κυρίου Κοσλόφσκι έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και αποσκοπούν ε, σε ε, καλύτερη διατύπωση και ελαφρά ε, διόρθωση των λεγόμενων της κυρίας Χίρσε. Θα ήθελε τελικά ο κύριος Κρουσόφσκι να ευχαριστήσει πολύ την κυρία Χίρσε ευελπιστώντας ότι θα δεχτεί τις τροπολογίες του. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του συναδέλφου Χέντελ, που είναι ασθενή σήμερα, λαμβάνω το λόγο γιατί είναι σκιώδη συγγετής για την ΚΟΥΑ για το θέμα αυτό και μου έχει σημειώσει ε, κάποιες παρατηρήσει. Καταρχήν, ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια, την κυρία Χίρς, για τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό. Δεν είναι απλό το θέμα αυτό ξέρουμε ότι είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και μεγαλύτερες αρμοδιότητες έχουν τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να τονίσουμε αυτά τα οποία μπορούμε για το έγγραφο της Επιτροπής για να μπορέσουμε να δώσουμε την απαραίτητη όθηση στις εργασίες αυτές πάντοτε την κριτική μας ε, την ε, ε, κάνουμε για να τονίσουμε ότι μιλάμε για την αγορά εργασίας περισσότερο παρά για την επαγγελματική κατάρτιση και μας ενδιαφέρει ε, να παίζει σημαντικό ρόλο ε, και ε, η κοινωνική προστασία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξουν κάποιες συμβιβαστικές λύσεις ακούγοντας ε, και τα όσα μας είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Ε, ο Τόμας Χέντελ εκ μέρους της ομάδας ε, της ΓΚΟΕ προτείνει τη βελτίωση της συνεργασίας και της συμμετοχής στο χώρο εργασίας και υπάρχουν αφορά έξι άρθρα, το 36, το 8, το 16 και το 23 μας ενδιαφέρει να τονίσουμε την ε, επαγγελματική κατάρτιση ε, και η αρμοδιότητα δεν θα πρέπει να είναι ε, μόνο αρμοδιότητα των εργαζομένων, αλλά θα πρέπει και η επιχείρηση ίδια να έχει κάποια ευθύνη για την κατάρτιση που θα πρέπει να παρέχει στους εργαζομένους. Και όσον αφορά την κοινωνική η ε, προστασία και ασφάλιση επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα θέματα. Μας ενδιαφέρει η έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ε, ε, σαν σύνολο και δεν θέλουμε με ένα κατακαιρματισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης ε, να χάνεται ε, η σημασία που παίζει η εκπαίδευση και κατάρτιση για τους ε, εργαζομένους και για τους νέους πιο συγκεκριμένα. Ακόμη κάποιες τροπολογίες ε, ίσως να πρέπει να δουλευτούν περισσότερο για να καταλήξουν ε, σε κάποια κοινή θέση μεταξύ των, ε, των ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Άντια Χίρς που είναι η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις. Κάποια σημεία τα έχουμε ήδη συζητήσει με τον κύριο Κοσλόφσκι για την σύνδεση που μπορεί να υπάρχει σε συγκεκριμένα σημεία. Ξέρω ποια είναι τα σημεία που θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικά. στις περισσότερες παρατηρήσεις νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ε, συνεννόηση. Ε, το θέμα του κατακαιρματισμού άκουσα πολλά επιχειρήματα. Υπάρχει δηλαδή ο φόβος ότι ε, η εκπαίδευση και κατάρτιση κατακαιρματίζεται ε, σε ενότητες μαθησιακές και έτσι θα χαθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καταλαβαίνουμε τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά παράλληλα υπάρχουν και ευκαιρίες που συνδέονται με τον διαχωρισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε modules. Βοηθάμε την κινητικότητα μέσα στην Ευρώπη κατά τον τρόπο αυτό και δίνεται η δυνατότητα να πάρει κανείς ε, το πτυχίο του σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα modules ε, της ενότητας κατάρτισης που λαμβάνει και σε άλλες χώρες, ούτως ώστε να μπορέσει κανείς ε, να βελτιώσει την κινητικότητα μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε αυτές ε, τις ε, ε, ανησυχίες. Και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένα σημαντικό θέμα. Δεν πρέπει να το δούμε μονομερός. Σε πολλούς τομείς υπάρχουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού και εδώ θα είχαν οι εργοδότες ακόμη μεγαλύτερο συμφέρον να υποστηρίξουν τους εργαζομένους να καταρτιστούν περισσότερο σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις. επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που θα μπορούσε να οδηγήσει τον εργαζόμενο και σε μια άλλη θέση εργασίας, σε μια άλλη επιχείρηση, σε ένα άλλο κλάδο. Πρέπει λοιπόν να το δούμε όχι μονομερός, αλλά και από την πλευρά του εργαζομένου και από την πλευρά του εργοδότου. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε με κάποιες συμβαστικές τροπολογίες ε, να καλύψουμε πολλές ε, προσδοκίες. Ευχαριστούμε πολύ την Άντια Χίους. 16 Μαρτίου ψηφίζεται στην Επιτροπή. Περνάμε τώρα στο σημείο που αρχικά θα έπρεπε να συζητηθεί πριν από την έκθεση τη Νάντια Χίξ είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κίνγκα Γκόντ. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση για την παράγραφο 9 αν καταλαβαίνω καλά για όλα τα άλλα θέματα, φαίνεται να έχουμε καταλήξει. Έχουμε συμβαστικές τροπολογίες, συμφωνούν όλοι από Συμφώνησε και το ΕΛΚΕ. ακριβώς έξω τώρα από την αίθουσα, αλλά εκρεμεί ένα θέμα και θέλω να σας περιγράψω πώς έχει η κατάσταση. Υπάρχει μία τροπολογία η οποία εκρεμεί. Δεν υπάρχει πλήρης ε, συμβιβασμός. Πρόκειται για την παράγραφο 9 όπως σας προείπα. Αυτό το οποίο εγώ λοιπόν προτείνω είναι ένα ταμείο το οποίο θα το διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μικρό ταμείο που θα έχει ωστόσο ακριβώς στόχο, ακριβώς αυτή της της και υπανάπτυκτες ε, κοινότητε. πέραν των ε, τρόπων ε, ε, διαχείρισης του κοινωνικού ταμείου και των άλλων ταμείων. Και στις προενταξιακές περιόδους η Κομισιόν είχε το καθήκον να διαχειρίζεται κάποια μικρά ταμεία τα οποία κατά κάποιο τρόπο είχαν συγκροτηθεί με βάση κάποιες καλές τοπικές πρωτοβουλίες και είχαν και ένα πιο μεγάλο χρονοδιάγραμμα για την υποστήριξη για μια βαθμιδόν προσέγγιση, μια σταδιακή προσέγγιση. Αλλά στην προτεξιακή περίοδο αυτό το οποίο το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι οι περισσότερες οργανώσεις, η τοπική κοινωνία, δηλαδή έμαθαν Πώ να κάνουν αιτήσει ε, χρηματοδότηση, επιχορήγηση, πώς να διαχειριστούν, έμαθαν λίγο τις γραφειοκρατικέ διαδικασίες, άρχισαν κατά κάποιο τρόπο να προσαρμόζονται στο σκέλος της μεταχρηματοδότησης, αλλά αυτές οι πάρα πολύ φτωχές κοινότητες ήταν απομονωμένες διότι ε, αν δεν υπήρχε απευθείας διαχείριση των ταμείων βάσει αυτής της αναπτυξιακής διάστασης, του αναπτυξιακού προσανατολισμού, δεν ήταν πρόθυμες ε, να ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει άμεση συμμετοχή των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Κάτι δηλαδή πρέπει να αντικαταστήσει τη γραφειοκρατία εάν θέλουμε να μειώσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η άμεση απευθεία συμμετοχή. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο προτείνω είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης αυτών των πολύ μικρής κλίμακας τοπικών πρωτοβουλειών που μπορούν αργότερα να μετεξελιχθούν σε πιο πολύπλοκα προγράμματα. Αυτή η άμεση συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχευση είπα, των, των πολύ καλών τοπικών πρωτοβουλειών με αναπτυξιακό προσανατολισμό είναι μια πρόταση, είμαστε εν μέσω αυτής της συζήτησης για το κατά πόσο θα υπάρχει αυτή η άμεση συμμετοχή για το κατά πόσο θα γίνει δεκτή ή όχι. Η εντύπωση που αποκόμισα και μετά από μακρά συζήτηση με κάποιε άλλε πολιτικέ ομάδε είναι ότι οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε είναι διατεθειμένε να στηρίξουν αυτή την προσέγγιση. Αλλά ακόμη μέσα σε διαπραγματεύσει με το ΕΛΚ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Και αν όχι θα δούμε ποια πρόταση μπορεί να στηριχθεί από την πλειοψηφία. Εγώ πάντως θα ήθελα να στηριχθεί η πρότασή μου. αλλιώ, και πάλι θα μείνουν εκτός αυτές οι κοινότητες. Και η χρηματοδότηση που είναι κατά κάποιο τρόπο προσανατολισμένη προ του Ρωμά δεν θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. στι πιο δηλαδή εξαθλειωμένε, πανάπτυκτε και απομονωμένε κοινότητε. Ευχαριστούμε. Cecilia Balsa Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέρντς για την ε, πολύ καλή δουλειά που έκανε για αυτήν την γνωμοδότηση. Ε, ένα κείμενο στο οποίο αναφέρονται τα πολύ απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε βελτίωση ε, την, τους Αθήγανους Ρωμά. Να ευχαριστήσω βεβαίως και την τους βοηθούς της κυρίας ε, Γκιόνες ε, που μας βοήθησαν πάρα πολύ και έδειξαν μεγάλη υπομονή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα ήθελα να καλέσω επίσης τους συναδέλφους να κατανοήσουν ότι ε, θα πρέπει οι πολιτικές προτάσεις να γίνουν με τρόπον ώστε να αναμειχθούν και οι ίδιοι οι Ρωμά στις αποφάσεις και στα μέτρα τα οποία θα ληφθούν επί τόπου προτάσεις οι οποίες θα αναγνωρίζουν επομένως και τον σημαντικό ρόλο των τοπικών κοινωνιών ε, και των τοπικών αρχών ε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως θα στηρίξει αυτές τις διαδικασίες. Σχετικά με τις τροπολογίες νομίζω ότι οι τροπολογίες είναι σωστές ε, γιατί συμπεριλαμβάνουν και την ανάγκη για προστασία και σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, για μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν απόρρια των επιτόπιων ερευνών, καθώς επίσης και και αναφέρουμε συγκεκριμένους τρόπους δράσης όπως αυτούς που ανέφερε και η συγγήτρια. Το σημαντικό είναι να φέρουμε τους Ρωμά μέσα στην κοινωνία όσον αφορά την τροπολογία 9. Το ζήτημα αυτό είμαι βεβαία ότι θα λυθεί ε, σήμερα και όχι αύριο και μια και είμαι και μέλος Επιτροπής ε, Ελευθεριών θα ήθελα να πω ότι θα προσπαθήσουμε και στην ε, άλλη Επιτροπή η εργασία να ε, συνεχιστεί κανονικά και να αντικατοπτριστούν στην έκθεση της ΛΥΜΠΕ όλα τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος και ο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί με πολύ σωστό τρόπο ε, έχει καταγράψει την έκθεση αυτή και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει είναι τα πλέον κρίσιμα. Πώς δηλαδή θα φτάσουν τελικά οι ευρωπαϊκοί πόροι εκεί που πρέπει και πώς θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς που πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί μέχρι τώρα δεν είδαμε και εξαιρετικές επιδόσεις. Άλλες χώρες τα χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά λάθος, άλλοι, ε, άλλες χώρες χρησιμοποίησαν τους πόρους αυτούς για άλλους λόγους και χάθηκαν εν ολίγης οι ευρωπαϊκοί πόροι σε όλους αυτούς τους δεδάλους. Η συγγήτρια ήταν πάντα στη διάθεσή μας, έδειξε μεγάλη διάθεση συμβιβασμού και πρέπει να πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς παρακολουθήσαμε την όλη διαδικασία γιατί θέλαμε μία έκθεση η οποία θα στηριχτεί από όλους. Το μόνο κρίσιμο και υποσυζήτηση ε, σημείο είναι αυτό της παραγράφου 9. Ενδεχομένως να παίζουν και κάποιο αρνητικό ρόλο οι ε, κακές μεταφράσεις του εγγράφου στις διάφορες ε, χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε άμεση σχέση ε, με την κοινωνία και με τις περιφέρειες. Απ' την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να επιβραδύνουμε τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κι άλλους οργανισμούς σε αυτήν την τόσο βραδικίνητη γραφειοκρατική Ευρώπη. Δεν θέλουμε ακόμα έναν οργανισμό που θα έχει ακόμα κάποια ε, ε, κάποιο περιεχόμενο εντολής και άλλωστε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν άμεση επαφή ανάμεσα στην Κομισιόν ε, και το την περιφέρεια. Αναρωτιέμαι, εάν αυτές οι κοινότητες Ρωμά είναι τόσο μικρές ε, και δεν έχουν καμία εκπροσώπηση, καμία, ε, ε, καμία οργάνωση, τότε ποιος θα μιλήσει εξ ονόματός τους, αν όχι η τοπική κοινωνία, οι τοπικές αρχές, μάλλον οι περιφερειακές αρχές. Με ποιον έχουμε άμεση επαφή, πώς γίνεται η άμεση επαφή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οργανώσεις. Επ' αυτού εμείς έχουμε κάποιους δισταγμούς και κάποιες αμφιβολίες. Και επομένως, χωρίς να θέλουμε να επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά ακόμα περισσότερο την σχέση ανάμεσα ε, στους τοπικούς πληθυσμούς και την Κομισιόν, θα πρέπει να βρούμε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου δεν θα δημιουργηθούν νέοι οργανισμοί αλλά ή να προβλέψουμε μια διατύπωση η οποία θα είναι πιο γενική, να αφήσουμε στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να παρέμβουν ακόμα και άμεσα στις μικρές κοινότητες Ρωμά και ας μην αποφασίσουμε από τώρα με συγκεκριμένο τρόπο για το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί η σχέση αυτή αργότερα θα μπορέσουμε ε, ε, σε συνεργασία και με τους οργανισμούς που δρούν επιτόπου θα μπορέσουμε λέω να ξανασυζητήσουμε το θέμα και να βρούμε ε, τις τελικές λύσεις. Δεν είναι ο σκοπός μας άλλωστε. Ο σκοπός της παρέμβασής μας είναι να δώσουμε στους Ρωμά την δυνατότητα να ενταχθούν γιατί να τους βοηθούμε διαρκώς χωρίς να τους κάνουμε τελικά να ενταχθούν δεν έχει έννοια. Έτσι διαβάζω εγώ αυτό το άρθρο και ελπίζω ότι εν τέλει θα βρεθεί μια λύση με την οποία θα ε, είμαστε σύμφωνοι όλοι. Ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ελπίζω να συνεισφέρετε στην εξέβρεση λύσεων. Η κυρία η επόμενη ομιλήτρια. Ε, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την υψηλή ποιότητα εργασία της. Το κείμενο το οποίο μας ε, προτείνει, το οποίο εμπλουτίζεται από πολύ σημαντικές τροπολογίες συμβιβασμού, δείχνει την σημασία του θέματος. Πρώτον να πούμε ότι η ένταξη των Ρωμά στην ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να περάσει από ένα πλέγμα ε, υπηρεσιών ε, καλής ε, ποιότητας από την ίδρευση μέχρι την αποχέτευση μέχρι την καλή στέγαση το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη την εκπαίδευση των παιδιών στην ουσία δηλαδή μέσα από το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεύτερον, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι ε, υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακριτική μεταχείριση η κοινότητα Ρωμά. Εκπροσωπούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρόλος μας είναι να αποφύγουμε τον στιγματισμό οποιασδήποτε κοινότητας. Δεν θέλουμε να στιγματίζεται λοιπόν η κοινότητα των Ρωμά. Ε, μέσα στην ε, διαφορά της εντάσσεται στην ευρωπαϊκή κληρονομιά και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Τέλος. Αναφέρεται στο κείμενο ότι οι πόροι βεβαίως θα πρέπει κατά προτεραιότητα να δίνονται στους Ρωμά. Μα γι' αυτό ακριβώς ε, ε, γράψαμε το κείμενο αυτό. Αυτό είναι ο ρόλος. Αλλά η διατύπωση δεν είναι ικανοποιητική. Και για να επανέλθουμε αυτήν την περίφημη τελευταία συμβαστική λύση. Πιστεύω ακράδαντα ότι όποια και αν είναι η διαδικασία θα πρέπει να ενταχθούν οι κοινότητες Ρωμά. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς τη θέση τους. Ε, θέλουμε να είμαστε κοντά τους, να κάνουμε πολιτική όχι για τους ανθρώπους, όχι για ε, τους πληθυσμούς αυτούς, αλλά μαζί τους, γιατί πολλές φορές έχουν εκείνη ήδη τις λύσεις. Δεύτερον, γίνεται λόγος για, μια ευρωπαϊκή, για ένα ευρωπαϊκό οργανισμό που θα διαχειρίζεται τους πόρους. Στην ουσία δεν είμαι κατά αυτής της ιδέας, είναι μια καλή ιδέα. Αλλά θα ήθελα να μάθω δύο πράγματα. Από τεχνικής απόψεως και από νομικής απόψεως. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Επίσης, ο οργανισμός αυτός, το ίδρυμα αυτό, ε, θα διαχειρίζεται και πόρους κοινωνικού ταμείου και ΦΕΝΤΕΡ. τότε είμαι απολύτως σύμφωνη. Άλλο ζήτημα. Θα πρέπει αυτός ο οργανισμός να εκπροσωπεί πραγματικά και την Ευρώπη και τους πληθυσμούς. Να μην παίρνει αποφάσεις η Ευρώπη ε, στην πλάτη τους, να μην παίρνει αποφάσεις η Ευρώπη για αυτούς ανταυτών. Και τέλος, ο ρόλος της διακυβέρνησης. Δηλαδή, αυτή η υπηρεσία, αυτός ο οργανισμός θα εργαστεί ε, σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό, ε, με την περιφέρεια, με ποιο βαθμό διακυβέρνησης θα συνεργαστεί. Και είμαι σίγουρη, είμαι βεβαία ότι θα βρούμε έναν πολύ καλό συμβιβασμό με την εισηγήτρια του θέματος αυτού. Ευχαριστούμε την Μαντελή και έχουμε ακόμη μία παρέμβαση. Ογκορεάνου. Ζητώ συγγνώμη για το πώς προφέρω το όνομά σας. Έχετε το λόγο. Καλή προσπάθεια πάντως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι νομίζω ότι η συγγήτρια με την οποία έχουμε έτσι, μια καλή παράδοση στο να συνεργαζόμαστε ωραία τα κατάφερε πολύ καλά. Θα έλεγα και εγώ ότι να είμαστε κοντά όπως είπε και η ίδια, όχι τόσο κοντά όμως. Παράγραφος 9. Είναι θέμα αρχής, αλλά και ουσίας. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και συγκεκριμένα τον κύριο Μπαλτασάρη που ανέφερε πάρα πολύ εύγλωτα την κατάσταση. Και πηγαίνω εγώ ακόμη πιο πέρα. Γιατί πρέπει να υποχωρήσουμε, να γυρίσουμε πίσω στην κατάσταση πριν την ένταξη. υπήρχαν οι μηχανισμοί που συγκροτήθηκαν τότε γιατί δεν υπήρχαν αυτοί που υπάρχουν τώρα. Γιατί να πάμε πίσω λοιπόν. Δεύτερον, πράγματι εγκυμονεί ένας πραγματικός κίνδυνος ε, γραφειοκρατικοποίησης του όλου πράγματος. Και υπάρχουν προβλήματα με τα χρήματα, τη χρηματοδότηση, πώς θα φτάσουν οι πόροι δηλαδή, τους πληθυσμούς ε, Ρωμά, τις κοινότητες Ρωμά, στην Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία. Υπάρχουν προβλήματα. Αλλά από τη δική μου εμπειρία και πώς να το θέσω. Επειδή υπάρχουν ε, κάποιες δυσλειτουργίες ε, και μπλοκαρίσματα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. η τοπική αυτοδιοίκηση σε μικρό επίπεδο μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη ευρωπαϊκή πολιτική να πάρει σάρκα και οστά, να γίνει μια τοπική πραγματικότητα. Διαφορετικά, φυσικά το να μιλάμε για δικαιώματα, για πρόσβαση των Ρωμά, Μπορούμε να κάνουμε τέτοιες πολύ γενναιόδορες ε, δηλώσεις αρχής, αλλά θα μείνουμε στα λόγια. Αυτό το οποίο λοιπόν ζητώ είναι να είμαστε πιο ρεαλιστές και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Και επανέρχομαι στην παράγραφο 9. Νομίζω ότι πρέπει να εμείνουμε σε αυτό το οποίο ε, έχουμε πει, να βελτιώσουμε αυτό που υπάρχει. Όχι ένας έξτρα μηχανισμός επίλυσης. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής που να ζητά το λόγο. Θα δώσω λοιπόν στην κυρία Κίνκα Γκόντ στην εισηγήτρια το λόγο για άλλη μια φορά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την τόσο ουσιαστική αυτή συζήτηση. Όπως βλέπετε όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και αυτοί που υπέβαλαν και συνέταξαν πολλές τροπολογίες ε, πραγματικά είναι αφοσιωμένοι, συμμετέχουν ε, βάσει της εμπειρίας τους. Και σίγουρα είμαι πεπισμένη ότι όλοι θέλουμε την καλύτερη δυνατή λύση και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι ναι μεν υπάρχουν συστήματα για την διάθεση πόρων στις χώρες αυτές και οι περισσότερες κοινότητες έχουν μάθει να αξιοποιούν και να χρησιμοποιούν τους σπόρους αυτούς. Και οι περισσότερες κοινότητες Ρωμά έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τους σπόρους αυτούς. Έχουν δηλαδή κάποια πρόσβαση στο κοινωνικό ταμείο, στα διαθροτικά ταμεία. Τώρα, δεν ξέρω ούτε κι εγώ αν είναι καλύτερη πρόταση αυτή που κάνω εγώ. Αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι πώς θα έχουμε πρόσβαση, πώς θα ε, προσεγγίσουμε αυτούς που είναι απομονωμένοι. Το είπε και ο κύριος Ε, δεν ψάχνουμε ε, πώς να σου το πω, ψάχνοντας κάποιους διάβλους, κάποιες άλλες εναλλακτικέ, εγώ σκεφτόμουν ε, πώς μπορούμε να φτάσουμε στις ε, απομονωμένες ε, πάμφτωχες κοινότητες που δεν έχουν πόρους. Και η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες χώρες υπάρχουν κάποια κομμάτια της κοινωνίας που έχουν μείνει εκτός και δεν αποφελούνται καθόλου από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συγκροτηθεί κάποιο καινούριο φορέα. Α μην κάνουμε τέτοια συζήτηση. Αυτό που ζητώ εγώ είναι η άμεση συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατάσταση της γραφειοκρατίας, αξιοποίηση της τοπικής γνώσης, των τοπικών διάβλων που υπάρχουν, που έχουν την εμπειρία, που έχουν τη γνώση και ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο αποδεκτό από όλους. Απλά θέλω να σας κάνω να καταλάβετε την πρωτοβουλία μου και πώς εγώ αντιλαμβάνομαι την κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, μπορούμε να ξανακαθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε να έχουμε ένα τελικό, ένα οριστικό κείμενο που θα μπορέσει να το στηρίξει η πλειοψηφία ή μακάρι να το στηρίξουν και όλες οι πολιτικές ομάδες γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Και πραγματικά με εξέπληξε και εμένα που για αυτό το τόσο μικρό κειμενάκι είχα σχεδόν 100 τροπολογίες να εξετάσω. Άρα καταλαβαίνω πόσο σημαντικό θεωρείτε και εσείς το ζήτημα αυτό και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ, Κίνγκα Γκέντς. Η ψηφοφορία είναι για αύριο. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα μπορέσετε να συμφωνήσετε για τα τελευταία ζητήματα που απομένουν. Δεν έχουμε άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Μπορούμε να τελειώσουμε λοιπόν λίγο νωρίτερα τη σημερινή μας συνεδρίαση. Αύριο να είμαστε εδώ στην ώρα μας στις 9 και θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Ασέια και θα είμαστε στη, στον τέταρτο όροφο, στην Αθουσα 1. Και θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Σάρι Εσαγιά για τις δημογραφικές αλλαγές και τις συνεπιές του στο μέλλον της πολιτικής συνοχής.